Good Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής μας. Όπως είπα προηγουμένως, συνεχίζουμε με τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας και καλωσορίζουμε τον Υπουργό κύριο Τομπίας, Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου της Σουηδίας. Το πρώτο που θα πρέπει να τονίσω είναι ότι τελευταία σκερούς όλο και περισσότερα μέλη ορίζουν στις κυβερνήσεις τους ειδικά υπουργό για αυτές τις πολιτικές πράγμα που αποδεικνύει πως η μετανάστευση και οι πολιτικές ασύλου και οι πολιτικές για τους προσφύγες είναι προτεραιότητες και στα εθνικά θεσμικά όργανα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από ευρωπαϊκής πλευράς υπάρχουν προτάσεις και πρωτοβουλίες νομοθετικές που πρόσφατα υπευλήθησαν στον τομέα αυτό και με τις οποίες θα ασχοληθούμε στην Επιτροπή μας. Αποτελούν μέρος του προγράμματος εργασίας του δικού μας. Μας απασχολεί κατά πρώτο λόγο λοιπόν αυτός ο πολλαπλασιασμός πρωτοβουλειών για να έχουμε μια προσέγγιση αποδοτική και συνεκτική, η οποία στα πλαίσια του προγράμματος της Στοκχόλμης θα ενδυναμωθεί. Γνωρίζουμε ότι η Υπουργό Μπέτρη Άσκ παρουσίασε και το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας και εμείς θέλουμε να υποβάλουμε συστάσεις για το θέμα αυτό για να βελτιωθεί και να ενισχυθεί το πρόγραμμα της Στοχόλμης, οι στόχοι του. Και κατά τη διάρκεια της δικής σας προεδρίας. Είμαστε πεπισμένοι ότι σύμφωνα με το πνεύμα και την διατύπωση της συνθήκης θα πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε στην εφαρμογή του προγράμματος Στοχόλμης κατά τη διάρκεια της ε, κοινοβουλευτικής μας θητείας που αρχίζει με την Σουηδική Προεδρία. Αυτή είναι μια δέσμευση που αναλάβαμε, την ε, εκφράσαμε την άποψή μας αυτή στην ε, κυρία Μπέτρις Άσκ και είπαμε ότι θα σας βοηθήσουμε κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας με τις συστάσεις και τα συμπεράσματα στα οποία θα καταλήξουμε σε εκθέσεις με τις οποίες θα ασχοληθούμε. Θα δώσω το λόγο στον Υπουργό κύριο Τομπίας γνωρίζοντας ότι πάρα πολλοί συνάδελφοι θα ζητήσουν να λάβουν το λόγο μετά από την παραβασή του. Θα ενεργήσουμε ως εξή. Θα έχουμε ένα πρώτο γύρο ερωτήσεων από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους της Επιτροπής, ώστε να ικανοποιήσω όλους τους συναδέλφους που θα θελήσουν να λάβουν το λόγο. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Το μικρόφωνο του Υπουργού παρακαλούμε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι και κυρίες βουλευτές. Είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα να εκπροσωπήσω την Σουηδική Προεδρία και να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Πολλές από τις απόψεις θα παρουσιάσω τις γνωρίζετε, κάποιες άλλες είναι νέες και θα ήθελα πριν αρχίσω πρώτα απ' όλα συγχαρώ διότι έχετε εκλεγεί μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις τελευταίες εκλογές και να συγχαρώ και τον πρόεδρο Λόπες Αγγιλάρ, τον πρόεδρό σας. Η Σουηδία συμμετείχε στις ευρωπαϊκές εκλογές του Ιουνίου με ποσοστό ανώτερο από αυτό του 2004 και είμαι πεπισμένος ότι από κοινού θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε σωστά και η υποστήριξη όλων των πολιτών προς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των θεσμικών οργάνων θα αυξήσει. Θα ήθελα αρχίζοντας να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης για μας και να αναφερθώ σε κάποια θέματα που αφορούν τη μετανάστευση και το άσυλο κυρίως να σας μιλήσω για την κατάσταση στη Μεσόγειο και για την παράνομη μεταναστή. Η συνάδελφός μου, η κυρία Άσκος, Υπουργός Δικαιοσύνης, ήδη σας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί και σας μίλησε για το στρατηγική που θα ακολουθούσουμε στα πλαίσια των θεμάτων της δικής της ευθύνης. Εγώ σήμερα το απόγευμα θα σας μιλήσω για τους στόχους μας, για τις φιλοδοξίες μας, για τις προτεραιότητές μας και να έχουμε μια Ευρώπη πιο ασφαλή και να εξασφαλίσουμε ίσα δικαιώματα σε όλους τους πολίτες. Σε θέματα μετανάστευσης έχουν γίνει μεγάλες εξελίξεις τα τελευταία χρόνια. Είδαμε πρόσφατα ότι υπάρχει νομοθεσία για μια κοινή πολιτική ασύλου και πολιτική μετανάστευσης. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία μελετούμε αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Τα κράτη-μέλη θέλουν να έχουν ένα σύστημα δικαιοσύνης δίκαιο και συνεκτικό για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και οι προκλήσεις της μετανάστευσης. Στα πλαίσια λοιπόν ενός συμφώνου μεταξύ των κρατών μελών θα ενισχυθεί αυτή η Επιτροπή. Στα πλαίσια της Επιτροπής Επίσης, υπάρχουν εξελίσεις, έχουν γίνει διάφορες διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, με τα διάφορα ε, εθνικά κοινοβούλια. Βλέπουμε ότι όλοι και περισσότερα πολίτες μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις που γίνονται για τη διαμόρφωση της, επιτροπή, της ε, πολιτικής μετανάστευσης. Έχουμε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ελευθερία και την Δικαιοσύνη που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο και η οποία ήδη παρουσιάστηκε στην άτυπη ε, συνεδρίαση των Υπουργών Δικαιοσύνης ε, στη Στοκχόλμη και Ξέρουμε ότι η κυρία Άσκ και ο κύριος Αγγιλάρ συμμετείχαν σε αυτήν την ε, άτυπη συνάντηση. Όπως είπε και η κυρία Άσκ, χρειάζεται καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών για να δούμε πώς θα ενεργήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε πάρα πολύ σωστά το πρόβλημα της μετανάστευσης για να είναι θετική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Θα πρέπει στα διάφορα κοινοβούλια τα, ε, να λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των κανόνων της χώρας προέλευσης και να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι οικονομικά εύρωστη για να μπορέσει να προσφέρει και απασχόληση στους οικονομικούς Επίση, Επίσης, ένα άλλο θέμα που μα απασχολεί είναι αυτό το θέμα τη δημοκρατική πρόκληση. Σήμερα διερχόμαστε όλοι μια περίοδο οικονομική κρίση, γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι μπορεί να κάνει το πρόγραμμα στους επόμενου μήνες, τα επόμενα χρόνια και να δούμε πώς οι διάφορες αλλαγές τα επόμενα πέντε χρόνια θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό αποτελεσματικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να προσελκύει εργατικό δυναμικό, να είναι οικονομικά ανταγωνιστική, αλλά θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της μετανάστευσης και να κάνουμε μια κοινή πολιτική. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις θετικές προκλήσεις της μετανάστευσης και να μπορέσουμε να δίνουμε οικονομικές και κοινωνικές λύσεις στους μετανάστες. Τα κράτη-μέλη από κοινού θα πρέπει να καταπολεμήσουν την παράνομη μετανάστευση και είναι σημαντικό να υπάρξει μια καλή ισορροπία μεταξύ των μέτρων ασφαλείας ώστε να μην δυσχεράνουμε υπερβολικά την νόμιμη μετανάστευση. Απ' την άλλη θα πρέπει να δούμε πώς θα ρυθμίσουμε το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών. Τα παιδιά που φτάνουν μόνα τους θα πρέπει να δούμε πώς θα τα υποδεχθούμε και θα τα βοηθήσουμε να ζήσουν καλύτερα. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν καλύτερο έλεγχο των μεταναστευτικών ε, ρευμάτων. Θα πρέπει να δούμε επίσης πώς θα καταμεριστούμε όλες τις ευθύνες. Οι μεταναστευτικές πιέσεις που ασκούνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με προσπάθειες που θα καταβάλουμε μακροπρόθεσμα, ώστε να μπορούμε να υποδεχόμεθα τους μετανάστες ή και κάποιους από αυτούς να τους επαναπατρίζουμε. Υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι πιο εκτεθειμένες σε αυτές τις μεταναστευτικές πιέσεις και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να υπάρχει κοινή πολιτική μετανάστευσης. Το σημείο κίνησης αυτής της πολιτικής θα πρέπει να είναι ε, υποδοχή των μεταναστών βάσει ε, των ιδίων κριτηρίων για όλους, κυρίως για τους ετούντες άσυλο. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μια πολιτική χορήγηση ασύλου πιο δίκαια και να επιτρέψουμε σε όλους να έχουν πρόσβαση σε αυτό το δικαίωμα αίτησης ασύλου βάσει δίκαιων κανόνων. Στα πλαίσια της Προεδρίας μας θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα και θα δούμε βάσει συγκεκριμένων δράσεων πώς θα ενεργήσουμε. Η Σουηδική Προεδρία έχει την πρόθεση να ενεργήσει με ανοιχτό πνεύμα, με διαφάνεια, ώστε τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη να ξέρουν τι ακριβώς κάνουμε. Στα πλαίσια του προγράμματος Στοκχόλμης Υπάρχουν κάποιες νομοθετικές δεσμεύσεις ε, τις οποίες έχουμε αναλάβει και θα θέλαμε να ακούσουμε και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάποιες επικοδομητικές προτάσεις τις οποίες ε, χρειαζόμαστε εάν θέλουμε να καταλήξουμε σε αποδοτικά και θετικά αποτελέσματα. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη έχει μεγάλες ευθύνες και αναλαμβάνει μεγάλες δεσμεύσεις σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας από κοινού και θα πρέπει να βασιζόμαστε σε μέτρα διαφανή, αντικειμενικά και απλά βάσει των διαφόρων συμβάσεων τους Γενέβης και άλλων οι οποίες αποτελούν την βάση του συστήματος ε, που μας επιτρέπει να δεχόμεθα μετανάστες και να χορηγούμε άσυλο. Ξέρουμε ότι κάποια κράτη-μέλη δεν μπορούν να οργανωθούν σε θέματα χορήγησης ασύλου, πράγμα το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις πολιτικές υποδοχής των ετούντων και ξέρουμε ότι πολλές φορές οι διαδικασίες είναι επαχθείς. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να, να καταβάλουμε προσπάθειες εναρμόνισης των μέτρων που ακολουθούμε. Η εργασία που επιτέλεσε η τσεχική προεδρία σε θέματα ασύλου ήταν εξαιρετική. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε και εμείς προσπάθειες για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το όλο σύστημα. Χρειαζόμαστε επίσης και την δική σας βοήθεια στο θέμα αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις και θα συνεχίσουμε την εξέταση των διαφόρων κεφαλαίων που αφορούν την πολιτική ασύλου για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε διάφορες νομοθετικές πράξεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στα διάφορα δίκαια στα πλαίσια καλής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Επίσης υπάρχουν διάφορα σχέδια για την εναρμόνιση και θα χρειαστούμε και πολύ καλή πρακτική συνεργασία, μάλλον σε πρακτικά θέματα μεταξύ όλων ημών. Ελπίζουμε ότι το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσουν σύντομα το φθινόπωρο να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία, δεδομένου ότι και για σας νομίζω ότι αυτό είναι θέμα προτεραιότητας. Την τελευταία Συμβούλιο Υπουργών αναφέρθηκε το θέμα της δημιουργίας μιας νέας επιτροπής, ενός νέου οργανισμού που θα χειρίζεται όλα τα θέματα ασύλου. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελπίζουμε ότι θα αποφασιστεί και θα ολοκληρωθεί ως το τέλος του χρόνου και ελπίζουμε ότι θα έχουμε ε, την συνδρομή υπαλλήλων που θα μας βοηθήσουν οι διάφοροι κανόνες που εφαρμόζονται για την πολιτική χορήγηση ασύλου να εφαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο και εναρμονισμένο ώστε να βοηθηθούν από την ύπαρξη αυτής της, αυτού του οργανισμού όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι το θέμα είναι αρκετά επίγον, δεν πρέπει να χάσουμε χρόνο. Ξέρουμε ότι έχουμε και τη δική σας υποστήριξη για το θέμα αυτό. Επίση, όσον αφορά τον κανονισμό Eurodac, Ελπίζουμε ότι μετά την κατάσταση τροπολογιών και τη συζήτηση θα μπορέσει να υπάρξει συμφωνία σε επίπεδο υπουργών. Υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις ακόμη, αλλά είναι προ συμφέρον όλων να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για αυτό τον κανονισμό Eurodac, ώστε να μπορέσει το σύστημα του Δουβλίνου να λειτουργήσει καλύτερα. Όσον αφορά τις ε, διάφορες συζητήσεις που θα γίνουν μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων, Ελπίζουμε ότι θα γίνουν σε πνεύμα θετικό και θα θέλαμε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταλήξουν σύντομα σε συμφωνία για το θέμα αυτό που να μπορέσει να ψηφιστεί σύντομα. Ελπίζουμε ότι τα μέτρα που προτείνει η Επιτροπή για τον Κανονισμό Eurodac θα μπορέσουν να εφαρμοστούν σύντομα. Θα ήθελα Επίσης, να βασιστούμε σε δουλειά που έχει επιτελεστεί στο παρελθόν για να προχωρήσουμε χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Όσον αφορά τις προτάσεις τροπολογιών για την οδηγία, για την υποδοχή, πρέπει να πούμε ότι η δική μας Προεδρία θέλει να εργαστεί και να συνεργαστεί στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Το Συμβούλιο πιστεύει ότι μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει περιθώριο ελιγμών και πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ θετικό να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσουμε σύντομα να καταλήξουμε βάσει αμοιβαίων συμβιβασμών και υποχωρήσεων σε συμφωνία. Σήμερα ε, βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο γίνονται επίκαιρα τα προβλήματα ασύλου. Υπάρχουν στην ε, περιοχή της Μεσογείου προβλήματα τα οποία μας αφορούν όλους και θα πρέπει να έχουμε μεγάλη ευαισθησία για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στις γειτονικές μας χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε την ε, παρούσα νομοθεσία, να μην φυστούμε προσπαθειών για να το κατορθώσουμε, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι νομοθετικές αλλαγές που θα γίνουν να έχουν σταθερές ε, βάσεις και να λάβουν υπόψη ότι πρέπει να γίνουν και μεγάλες χρηματικές προσπάθειες στα κράτη της Μεσογείου. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολλοί σαφείς πολιτικές συμφωνίες για να ολοκληρωθούν αυτές οι πολιτικές. Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου που θα θέσουμε σε το αργότερο το 2010. Τελικός, ε, τελική, το πρόγραμμα της Χάγης κατέληξε σε κάποιες νομικές προτάσεις και σε κάποια μέτρα τα οποία θα πρέπει να μας βοηθήσουν να χειριστούμε το πρόβλημα της χορήγησης ασύλου με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει και να τις ολοκληρώσουμε. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό και επαναλαμβάνω θα πρέπει να έχουμε και την δική σας υποστήριξη στο Συμβούλιο. Ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά άτομα ε, χρειάζονται προστασία και υποστήριξη, αλλά και σε άλλες περιοχές του κόσμου έχουμε στρατόπεδα στα οποία ζουν πρόσφυγες σε πολύ πρόσκαιρες συνθήκες και πρέπει να τα βοηθήσουμε να βελτιώσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκουμε. Ένα πολύ σημαντικό θέμα στα πλαίσια πολιτικής ασύλου είναι να λαμβάνουμε υπόψη την εξωτερική διάσταση αυτής της πολιτικής ασύλου την οποία θέλουμε να δημιουργήσουμε. Αυτό είναι και για μας προτεραιότητα. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι με μεγάλη ευχαρίστηση σα υποβάλλω αυτέ τι προτάσει και να σα πω ότι με μεγάλο ενθουσιασμό εργαζόμαστε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σύντομα σε πολιτική συμφωνία. Η κατάσταση στη Μεσόγειο αποδεικνύει με σαφήνεια ότι χρειαζόμαστε μια συγκεκριμένη πολιτική μετανάστευση και ασύλου. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τους ε, ε συνδρομή σας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε τα πλαίσια του Συμβουλίου σε κοινή πρωτοβουλία που θα περιλαμβάνει όλη τη λεκάνη του, της Μεσογείου. Καθώς και για τη συνδρομή σας για άλλες ε, στρατηγικές πρωτοβουλίες. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω Καταλαβαίνω τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μάλτα, η Κύπρος, η Ιταλία και η Ελλάδα. Πράγμα που σημαίνει ότι απαιτούνται ειδικά μέτρα για να μπορέσουν να αμβληνθούν οι πιέσει από τα μέσα συγγνώμη, ρεύματα που ασκούνται στι χώρε αυτέ. Η Συνδική Προεδρία θα ήθελε να πει ότι θα θέλαμε να υπάρχει επικοδομητική στάση εκ μέρους όλων ώστε όλοι μαζί στην ΚΝΟΥΡ, στην Frontex, εσείς και εμείς να βρούμε πώς θα μπορέσουμε να λύσουμε μακροπρόθεσμα το πρόβλημα αυτό της μετανάστευσης που πιέζει, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα στις χώρες της Μεσογείου. Κυρίες και κύριοι, είναι πολύ σημαντικές οι σχέσεις μας με τα άτομα τα οποία ζουν και εντός και εκτός κοινότητες και που θέλουν να εργαστούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μετακομίσουν στις χώρες μας. Θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή πολιτική μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις αυτών των ατόμων. Και θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχουν ε, αναλυφθεί για αυτό το, αυτό το θέμα. και να συζητήσουμε και να επιλύσουμε επίσης το θέμα των θεωρήσεων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ξέρουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, ταχύτητες που μπορούν να ακολουθούν μεταξύ των διαφόρων χωρών της περιοχής αυτής. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε ε, να διευθετήσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Επίσης υπάρχουν ε, θα είναι ένα θετικό μήνυμα αυτό προς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, εάν δηλαδή ε, τους δοθεί απαλλαγή από την ε, ε, υποχρέωση να λαμβάνουν προξενικές θεωρήσεις και θα είναι θετικό όπως λέω το μήνυμα. Θα αναμείνουμε τώρα όμως και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όπως και η Τσεχική Προεδρία θα συνεχίσουμε με το πρόβλημα πληροφοριών για προξενικές θεωρήσεις. Τον Δεκέμβριο ακόμα το σύστημα δεν θα είναι λειτουργικό λόγω τεχνικού προβλήματος, ενώ έτσι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Όμως δεν επιτρέπεται να καθυστερήσει περισσότερο η έναρξη της φάσης λειτουργίας. Στο μεταξύ πάντως διευκολύνεται η, ε, η δυνατότητα κατάθεσης αιτήσεων για προξενικές θεωρήσεις με βιομετρικά δεδομένα και ούτω καθεξής. Και θα είναι από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την κοινή πολιτική προξενικών θεωρήσεων. Ιδού λοιπόν οι βασικές γραμμές της ε, Προεδρίας και αναμένω βεβαίως με ενδιαφέρον την ε, συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μεταξύ είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είμαι βέβαιος ότι μπορεί να αρχίσει τώρα η συζήτηση. Όπως είπα, προτείνω να περιοριστούμε σε ό,τι αφορά το χρόνο αγορεύσεως, ώστε να μπορέσουν να λάβουν όσο το δυνατόν περισσότεροι βουλευτέ τον λόγο. Έχουμε σημειώσει ήδη εκτό των συντονιστών των ε, πολιτικών ομάδων. Έχουμε λοιπόν σημειώσει άλλα 15 ονόματα. Α, ακόμη ένα όνομα, Κέλλερ. Α, Κέλλερ περιλαμβάνεται μεταξύ των 15 ονομάτων. Ε, και ο κύριος Μαστέλα. Λοιπόν, προτείνω τώρα να ε, κλείσουμε τον κατάλογο των αγορητών, διότι έτσι δεν θα προλάβουμε. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα λοιπόν να ε, σεβαστείτε τον περιορισμό χρόνου. Έχει καλώς. Λοιπόν, δίνουμε τώρα τον λόγο πρώτα στον κύριο Μπουσούτιλ, εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίαση εξ ονόματος της ομάδας του Λαϊκού Κόμματος σας διαβεβαιώ για το ανοιχτό πνεύμα με το οποίο θα προσεγγίσουμε την συνεργασία μαζί σας ε, τους επόμενους μήνες για να σας ε, βοηθήσουμε να επιτύχετε τους στόχους σας σε αυτό τον αμφιλεγόμενο και δύσκολο, περίπλοκο τομέα της εξωτερικής πολιτικής που ωστόσο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί ε, σημαίνονται πολλές εξελίξεις και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πολλά πράγματα συμβαίνουν και επιτόπου. Και όχι μόνο επιτόπου, αλλά και στην θάλασσα. Η χώρα μου, η Μάλτα, αυτή τη στιγμή επιτρέπει την ε, προσέγγιση στις ε, ακτές της ε, μίας λέμβου με 85 πρόσφυγες οι οποίοι διεσώθηκαν πριν από λίγα ε, πριν από λίγη ώρα από ε, ένα σημείο περίπου 85 μίλια από την Λαμπεντούσα. Αυτό που χρειάζεται είναι η κοινή επικοδομητική λογική που πρέπει να εμπνεύσει τις συζητήσεις, τις συζητήσεις μας. Διότι οι πολίτες ρωτούν, μα τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά επιτέλους πόσο αποτελεσματική είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Και θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί όταν απαντούμε στις ερωτήσεις αυτές. Η απάντηση που δίνω εγώ είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά αποτελεσματική. Δεν είναι καθόλου αποτελεσματική. Γι' αυτό και απαιτείται η δική σας σύμβολη. Μίλησατε για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Σας διαβεβαιούμε ότι θα συνεργαστούμε μαζί σας για να συμβάλλουμε στην επίτευξη των στόχων σας. Αυτά όμως είναι τα σχέδια για την επόμενη πενταετία. Αυτό που μας απασχολεί εμάς εδώ και σήμερα είναι πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ώστε τα όσα έχουμε ήδη συμφωνήσει όπως το πακέτο μεταναστεύσεως και ασύλου του περασμένου Οκτωβρίου, πώς αυτά θα εφαρμοστούν. Εδώ έχουμε αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των ήδη συμφωνηθέντων σύντομα τέσσερα σημεία όπου θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση για να εξασφαλιστεί επαρκής εφαρμογή των ε, συμφωνηθέντων. Πρώτο, η ανάγκη να συνεχιστεί η ε, μάχη, ο αγώνας κατά της παράνομης μετανάστευσης. Είτε το θέλουμε είτε όχι, οι διαδρομές που ακολουθούν οι μεταναστεύσεις ε, στη Μεσόγειο είναι παράνομες και πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την νόμιμη μετανάστευση. Μιλώ για παράνομη μετανάστευση. Και εκεί αυτήν πρέπει να την σταματήσουμε. Για να μπορέσει να γίνει αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι θα σταματήσουμε και τις ανθρώπινες τραγωδίες που σημειώνονται. Ενίσχυση λοιπόν πρώτα της Frontex. Ενίσχυση των προσπάθειών μας για συντονισμένες ε, προσπάθειες, πρωτοβουλίες επιστροφής των προσώπων αυτών στις χώρες προέλευσης τους. Εάν λοιπόν δεν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες και κυρίως τις χώρες προελεύσεως, αλλά και ορισμένες χώρες διαμετακομίσεως, διελεύσεως, δεν θα μπορέσουμε να σταματήσουμε την ιστορία αυτή. Στην Μεσόγειο είναι σαφές ότι εάν δεν εξασφαλίσουμε τη συνεργασία χωρών όπως η Λιβύη, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ανακόψουμε τις παράνομες οδούς μεταναστεύσεως. Δεύτερο, ο πρόεδρος, ναι, ναι παρακαλώ ολοκληρώστε κύριε Μπουσούτη. Ορισμένες χώρες μέλη, κυρίως οι νότιες χώρες μέλη, ζητούν μηχανισμούς αλληλεγγύης. Θα αναμείνουμε να ακούσουμε με ενδιαφέρον τι έχετε να πείτε σχετικά. Τέλος, το ε, γραφείο υποστήριξης, το Ευρωπαϊκό Γραφείο υποστήριξη Ασύλου. Εμείς ενδιαφερόμαστε πολύ να συνεργαστούμε και θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί σχετικά σύντομα μια συμφωνία. Σας ευχαριστώ κύριε ε, Υπουργέ. Ο κύριος Μωράης παρακαλώ σεβαστεί το όριο των τριών λεπτών. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Όπως και η Φιλανδική Προεδρία Προδεκαετία, νομίζω και η δική σας κάνει σημαντική προσπάθεια για τη δημιουργία μιας κοινή πολιτικής ασύλου. Όμως αυτό είναι και το πρόβλημα. Σας ρωτώ και εγώ, όπως ο προηγούμενος, τι ε, έχετε να πείτε σχετικά με τις προσωρινές προτάσεις. Έχει παρέλθει μια δεκαετία. Έκτοτε και ακόμα δεν έχουμε την κοινή πολιτική ασύλου. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεστε να αναλάβετε και ποια είναι η προοπτική που δίνεται σχετικά με, τον, μια ρεαλιστική, εν πάση περιπτώσει, προοπτική για την κοινή πολιτική ασύλου. Το θέμα είναι περίπλοκο βέβαια. Καλωσορίζουμε επίσης το γεγονός ότι έχει γίνει πολλή δουλειά στην προηγούμενη θητεία του Κοινοβουλίου για το πακέτο του ασύλου. Και κυρίως για το Γραφείο Υποστήριξης ε, Ασύλου. βασίζεστε σε αυτά που έχει ε, εγκρίνει το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία και που ήταν προϊόν ε, προσεκτικής διαβούλευσης. Και η έκθεση του Αντώνιο Μάσεν Πιτάργου που περιέλαβε σημαντικές βασικές αρχές που να καταστήσουν μια κοινή, ενδεχόμενη κοινή πολιτική ασύλου ισορροπημένη. Όπως είπε και ο κύριος Μπουσούτιλ, από αυτά πλήττονται κυρίω οι νότιε χώρε. Οποιαδήποτε κοινή πολιτική ασύλου θα πρέπει να είναι περιεκτική. Και η πολιτική του Τάμπερε τότε είχε ε, αυτό το όραμα. Πώ βλέπετε το όραμα εκείνο του 1999 και πώ βλέπετε την προοπτική τώρα. Χάρηκα για το όσα είπατε για το πακέτο του ασύλου και θα αρκεστώ σε αυτά τα σχόλια. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ενίς Πλασάρτ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Είχαμε, είχα τη δυνατότητα να σήμερα σύντομα μαζί του και διαπίστωσα ότι και, ε, τα, τα, σχέδια της, της Ιουδικής θα, υποστηριχθούν από την πολιτική μας ομάδα. Ορισμένα από τα οποία είπε ο κ. Μπουσούτιλ με βρίσκουν σύμφωνοι. Δηλαδή η έλλειψη αλληλεγγύης, μεταξύ των χωρών μελών αποτελεί όντως ένα εμπόδιο για την καθίδρυση μιας κοινή πολιτικής ασύλου. Και εξετάζοντας την συνοφορά της ε, Frontex την εμπειρογνωμοσύνη που συλλέγεται, βλέπετε ποιε είναι οι χώρε που είναι στην πρωτοπορία και αυτέ είναι που καλούνται, προ την πρώτη γραμμή μάλλον, και αυτέ είναι που καλούνται εν τέλει να πληρώσουν τα σπασμένα. Ο βολονταρισμός δεν πρόκειται να οδηγήσει σε λύσεις τις χώρες μέλη σε θέματα όπως της επανεγκατάστασης ε, παράνομων μεταναστών. Το Κοινοβουλίο στην προηγούμενη θητεία του βέβαια είπε ότι δεν μπορεί να είναι εθελοντική συμμόρφωση η συμφωνία, θα πρέπει να είναι υποχρεωτική. Κάθε χώρα θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της. Θα πρέπει να ληφθούν λοιπόν δεσμευτικά μέτρα ε, για να αναγκάσουν τις χώρες να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ελπίζω η ε, ε, Σουηδική Προεδρία να τα καταφέρει και κυρίως με τις διμερεί σχέσεις της με τις ε, χώρες μέλη. κυρία θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία ενός υπουργού μιας χώρας η οποία υποστηρίζει το μεγαλύτερο αριθμό και δέχτηκε στη χώρα του Ιρακινούς πρόσφυγες. Είναι μια ηγετική θέση την οποία έχετε και νομιμοποιεί και τις προτάσεις σας άλλωστε, η στάση σας αυτή. Σχετικά με τις διαπραγματεύσεις τις οποίες ελπίζει να ολοκληρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε επαφές αναφέρομαι με τη Λιβύη για την υπογραφή μια συμφωνία συνεργασίας η οποία θα καλύπτει και τις μεταναστευτικές ροές. Τίθενται ορισμένα ερωτήματα τα σχετικά με τα δικαιώματα των μεταναστών και τη μη παραβίαση της αρχής της C'est-à-dire le fait qu'elle renvoie des personnes qui sont éventuellement en demande de protection internationale, qui sont renvoyées et ça a été condamné. Της αρχής της επαναπρόθεσης λοιπόν. Η στάση χωρών όπως η Ιταλία έχει καταδικαστεί από πολλές άλλες χώρες, από το Συμβούλιο της Ευρώπης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα είναι ότι δημιουργείται κίνδυνος για πάρα πολλές χώρες ε, να τύχουν κακής μεταχείρισης. Έχω επισκεφθεί μαζί με τον κύριο Μπουσούτιλ ένα κέντρο κράτησης μεταναστών στη Λιβύη και διαρωτώ με για το τι εννοούμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όταν λέμε ότι θέλουμε εγγυήσεις έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά και βρίσκονται στη Γαλλία σαν παράδειγμα και ε, επιστρέφουν στη Λιβύη, πώς θα αντιμετωπιστούν με ε, ανθρώπινο τρόπο και πώς μπορούμε εμείς να αξιολογήσουμε την κατάσταση αυτή λόγω των επιπέδων δημοκρατίας που υπάρχουν στη χώρα αυτή και στην ανυπαρξία ουσιαστικά της κοινωνίας των πολιτών. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι θέλετε να καταστήσετε αρκετά αποτελεσματικότερα από ό,τι σήμερα τα συμπεφωνημένα στο Δουβλίνο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να διαγραφούν τα συμπεράσματα του ε, Δουβλίνου για τρεις λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι αν πράγματι επιθυμούμε και νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος ενός κοινού καθεστώτος ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον θέλουμε λοιπόν είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ορίσουμε τα κατάλληλα επίπεδα προστασίας έτσι ώστε τα πρόσωπα αυτά, τα υποψήφια, να επιλέγουν τις χώρες στις οποίες έχουν τις περισσότερες δυνατότητες. Η συμφωνία του Δουβλίνου όμως δεν το επιτρέπει κάτι τέτοιο, υποχρεωτικά μένετε στην πρώτη χώρα στην οποία πηγαίνετε, χώρα στην οποία ίσως να μην έχετε κάποιους δεσμούς ιστορικούς, οικογενειακούς, οικονομικούς ή οτιδήποτε άλλο. Δεύτερον, αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν σε μια χώρα της Ευρώπης ε, δεν τολμούν να διεκδικήσουν χορήγηση ασύλου, γιατί φοβούνται ότι θα σταλούν σε μια χώρα σαν την Ελλάδα όπου δεν υπάρχει καμία δυνατότητα και είναι ένα πραγματικό εμπόδιο στην διεθνή προστασία η στάση τέτοιων χωρών. Και η τρίτη περίπτωση και ο τρίτος λόγος αν θέλετε που γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνες, Ιταλοί και Μαλτέζοι συνάδελφοι είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και δεν μπορούν να γίνουν ε, αντικείμενο σωστής διαχείρισης. Παρακαλώ να τελειώνετε λέει ο Πρόεδρος. Πώς λοιπόν θα απαντήσετε παρακαλώ σε αυτές τις τρεις ε, βλαβερές συνέπειες των συμφωνιών του Δουβλίνου σήμερα. Ο κύριος Κίρκοπφ. Ζητώ συγγνώμη γιατί δεν άκουσα όλες τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Σαν τέος υπουργό Μετανάστευσης του Ηνωμένου Βασιλείου ε, γνωρίζω τις ε, ε, προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει και αυτό στη χώρα του. Παρ' όλα αυτά έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει να είμαστε <clears throat> Ε, να γνωρίζουμε το πρόβλημα και να προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε λίγο τα θέματα της μετανάστευσης από τη μία και του ασύλου από την άλλη. Σαν δικηγόρος γνωρίζω ότι οι κανόνες είναι κανόνες και οι κανόνες για τη μετανάστευση θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί και υπάρχουν τα εθνικά συμφέροντα και οι προτεραιότητες της κάθε χώρας είναι αυτές που καλύπτει τις οικές της ανάγκες. Για την μετανάστευση τώρα αυτά για, την, για το άσυλο. Φαίνεται ότι έχουμε ένα πρόβλημα εδώ. Το άσυλο χρησιμοποιείται πάρα πολύ συχνά για καταχρηστική θα έλεγα υπερκέραση του ε, κανονικού δικτύου το οποίο καλύπτει τα θέματα της μετανάστευσης. Νομίζω ότι δεν έχω να προσθέσω πολύ περισσότερα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πιο αυστηροί, να συνεργαστούμε σωστά και να αντιμετωπίσουμε αυτές τις χώρες που ενθαρρύνουν ουσιαστικά τους κατοίκους τους να έρθουν στην Ευρώπη Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις αντιμετωπίζουν τρομερούς κινδύνους όταν ταξιδεύουν προς την Ευρώπη και τρομερούς κινδύνους όταν είναι στην ίδια την Ευρώπη. Οι χώρες αντιληβή υποστηρίζουν πρακτικές που πιέζουν την Ευρώπη με απαράδεκτο τρόπο και μάλιστα οι πρακτικές αυτές είναι απαράδεκτες και για τους ίδιους τους υποψήφιους μετανάστες. Οι απώλειες ζωής στην ανοιχτή θάλασσα είναι φρικτές ε, σαν συνθήκες θα έλεγα. Συνεπώς θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες ε, της Ευρώπης που δεν έχουν ε, τους πόρους τους οποίους έχουν ανάγκη και που έχουν να αντιμετωπίσουν στην περιφέρεια της Ευρώπης με μια υπερβολική πίεση ε, και εμείς δεν θα πρέπει να κρύβουμε το πρόβλημα, δεν θα πρέπει να μην τους βοηθάμε, αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα τα δικαιώματα των κρατών μελών να εντάσσουν στους κανόνες τους τις βασικές τους προτεραιότητες. Κύριος Ταβάρες. Χαίρετε κύριε Υπουργέ. Χαίρετε αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζοντας θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά την παράνομη μετανάστευση, το πρόβλημα πολλές φορές τίθεται με ασφαλμένο τρόπο. Οι μετανάστες που φάνουν από τις νότιες χώρες στην Ευρώπη είναι σε μεγάλο βαθμό όσοι φτάνουν από την Αφρική μέσω της Λιβύης είναι άτομα που ζητούν άσυλο και πολλές φορές έχουν το δικαίωμα και κατορθώνουν να πάρουν και το άσυλο σε ευρωπαϊκές χώρες. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα παράνομων δρόμων, αλλά πώς θα μπορέσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές ασύλου να τις προσαρμόσουμε με τρόπο ώστε να γίνεται η αίτηση και η χορήγηση του ασύλου με, ασφα... με συνδίκες ασφαλείας για τα άτομα τα οποία το δικαιούνται όταν το ζητούν το άσυλο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε την εντολή που έχει δοθεί στην Frontex ώστε να λαμβάνεται υπόψη αυτό το δικαίωμα που έχουν οι ετούντες άσυλο. Θα πρέπει επίσης να πω ότι είπαμε ότι θα πρέπει εδώ να κάνουμε κάτι κατά των παράνομων ε, οδών ε, μετανάστευσης. Εντάξει, σωστό και λογικό. Κάτι που είναι παράνομο πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Βεβαίω είναι εύκολο να το λέμε στα λόγια, αλλά είναι πολύ δύσκολο στα έργα να το κάνουμε αυτό και στην πράξη. Τι συμβαίνει λοιπόν. Κινδυνεύουμε να εμπλακούμε σε μία μαξιμαλιστική και μη ρεαλιστική πολιτική όσον αφορά το στόχο. Άρα, μια πολιτική η οποία είναι καταδικασμένη να ε, αποτύχει. Όπως και άλλες πολιτικές. Πολλές φορές είναι ρητορικές, εσφαλμένες, αλλά δεν έχουν καμία πρακτική αξία. Θα είναι λοιπόν εύκολο μετά να ε, εκφράζει κανείς τη λύπη του, διότι δεν μπόρεσε να υπάρξει σωστή πολιτική και αλληλεγγύη για να καταπολεμηθούν αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν η Σουηδική Προεδρία να μπορέσει να σκεφτεί πάρα πολύ σωστά αυτό το θέμα της πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου για να μπορέσει να κάνει μια πολιτική ρεαλιστική. Διότι οι μη ρεαλιστικές πολιτικές, επαναλαμβάνω, μπορούν ώρες-ώρες να οδηγήσουν και σε... Ε, πολιτικές που διέπονται από ανήθικες αρχές. Πολιτικές που οδηγούν στο θάνατο των ατόμων που ζητούν άσυλο, στη θάλασσα. Πώς κατέληξαν εκεί. Πολλές φορές αυτό το πρακτικό αποτέλεσμα εδράζεται σε εσφαλμένες πολιτικές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποργέτσιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η νομιμότητα είναι ένα θέμα για το οποίο κανείς δεν αμφιβάλλει. Υπάρχουν άτομα τα οποία δικαιούνται να ζητήσουν άσυλο αλλά αυτό δεν δικαιολογεί τις ύπαρξη μη πολιτικής ή μια πολιτική που θα τους ε, οδηγήσει σε μια πιο δύσκολη κατάσταση. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω την παράνομη μετανάστευση την οποία χειρίζονται πολλές φορές μαφιόζοι. Ή ακόμη και τρομοκράτες. Θα πρέπει λοιπόν αυτά το θέμα να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Κύριε Υπουργέ, αναφέρατε αυτά τα θέματα κάπως ακροθυγός. Γι' αυτό θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με τους συναδέλφους που είπαν ότι θα πρέπει η Ευρώπη να αναλάβει δεσμεύσεις για να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση, αλλά και να κάνει κάτι για να προληπτικά, να προλάβει τέτοιου είδους καταστάση. Επίσης, οι χώροι διέλευσης, οι περιοχές διέλευσης θα πρέπει να την χάνουν καλύτερο ελέγχου. Υπάρχουν χώρες διέλευσης από τις οποίες φτάνουν οι μετανάστες τι έκανε όμω η Ευρώπη στι χώρες της Αφρική από τις οποίες φτάνουν όλα αυτά τα μεταναστευτικά παρανομαρεύματα. Τι έχει κάνει για να μπορέσει κατά κάποιο τρόπο εκεί όπου γίνεται και εμπορία ατόμων από αυτού που οδηγούν του λαθρομετανάστες στι πόρτες μας ε, ώστε να μπορέσει να καταπολυθεί αυτό το φαινόμενο. Είναι λοιπόν απαραίτητο και σημαντικό να βοηθηθούν και αυτές ε, οι χώρες που βρίσκονται στην προμετωπίδα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Και βεβαίως θα πρέπει να έχουμε πολιτική επαναπροώθηση των μεταναστών, αλλά θα πρέπει να έχουμε και μια πολιτική βοήθειας των χωρών που υποφέρουν ε, από αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα. Πρέπει να πω ότι εκτός από τις ε, ατέρμονες συζητήσεις που κάνουμε, θα πρέπει να κάνουμε και κάτι το σημαντικό και συγκεκριμένο, όπως έκανε και η δική μας, το δικό μας ε, Ιταλικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, ακούσατε τις παρατηρήσεις, τις δικές μας, τις παρατηρήσεις των συντονιστών και μπορείτε να απαντήσετε για να αρχίσουμε μετά την κανονική συζήτηση με τα άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τα ενδιαφέροντα σχόλια. Θα αρχίσω με αυτό του κυρίου Μπούσουτιλ. Είναι σημαντικό όντως να τονίσουμε την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα του η Μάλτα. Προσωπικά επισκέφθηκα την Μάλτα στις αρχές του καλοκαιριού για να δω τα πράγματα επιτόπου. Σημειώνω ότι είναι όντως ιδιαίτερα σημαντικό να εξετάσουμε το θέμα ρεαλιστικά. Δεν είναι δυνατόν να δοθούν πρόχειρες λύσεις σε θέματα μετανάστευσης. Να βελτιώσουμε το σύστημα ασύλου, αλλά ταυτόχρονα να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε έναν ξεκάθαρο, ανοιχτό διάλογο με, τρεις, με, με, τρίτες χώρες. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια επίλυση του προβλήματος. κυρία Φλότρα είπε επίσης Ανέφερε επίση το πρόβλημα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και Λιβύης. Τονίζω ότι με συζητήσεις για, σχετικά με μια συμφωνία πλαίσιο με τη Λιβύη αποτελούν το κλειδί για την πρόοδο. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μπαρό θα επισκεφθεί Τουρκία και Λιβύη στη διάρκεια του φθινοπόρου. Ε, πιστεύω ότι αυτή η επίσκεψη μπορεί να βοηθήσει διότι δείχνει ότι έχουμε εν τέλει επαφές με τρίτες χώρες όταν πρόκειται για θέματα μεταναστεύσεως, για την ανάπτυξη ικανοτήτων αντιμετώπιση του προβλήματος, ε, για την προστασία εν τέλει των ανθρώπων. Πάντως πρέπει να διασφαλίσουμε τη σωστή χρήση των μέσων που διαθέτουμε. Για παράδειγμα, η εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει ο Ήπατος αρμοστή για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ. Αυτά μας χρειάζονται και να μπορούμε να βασιστούμε σε αυτή την εμπειρογνωμοσύνη όταν συζητούμε με Τουρκία και Λιβύη. Η σημασία της νόμιμης μετανάστευση είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλη. Η παράνομη μετανάστευση είναι ο μεγαλύτερο εχθρό τη νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει προσπαθώντας να αντιμετωπίσουμε την μία, την παράνομη δηλαδή, να ε, ρυθμίσουμε και τα της νόμιμης μετανάστευση Εμείς θεωρούμε στην Στοκχόλμη ότι αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Μωράες. Μιλήσατε για το στρατηγικό υπόβαθρο. Το όραμα του Τάμπερε θα συνεχίσει να ζει και μέσα στα πλαίσια του προγράμματος της Στοκχόλμης. η αναζήτηση της ισορροπίας αυτής μεταξύ των υποχρεώσεων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει τα σύνορά της από την μεριά και από την άλλη να είναι ανοιχτή απέναντι στον υπόλοιπο κόσμο είναι κάτι που η Ασυρική Προεδρία το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Η κυρία Ενής Πλαθκάρτ. Όντως υπήρξε έλλειψη αλληλεγγύης έλλειψη ε, μιας προσπάθειας ανάληψης των βαρών και των ε, ευθυνών, αλλά πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Ο κ. Κέρκο βεβαίω έχει δίκιο στα όσα επισήμανε για τη μετανάστευση και το άσυλο. Το άσυλο είναι δικαίωμα των ανθρώπων, ενώ η μετανάστευση είναι ζήτημα δυνατοτήτων. Όταν μιλούμε για νόμιμη μετανάστευση προς την Ευρώπη και επιθυμούμε να ρυθμίσουμε τα σχετικά, αυτό θα πρέπει να γίνει στη βάση των αναγκών, των υφισταμένων αναγκών. Θα πρέπει οι χώρες μέλη να μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το ύψος, με τον αριθμό των ε, μεταναστών που μπορούν να υποδεχθούν. Το ίδιο για το άσυλο. Και αυτά θα περιληφθούν στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Για τον κύριο Ταβάρες, η συστηματική εφαρμογή του κοινού συστήματος ασύλου. Έχουμε την καταρχήν πολιτική συμφωνία, διαθέτουμε τη σχετική νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποσύσει τις ευθύνες της επί του προκειμένου, εφόσον ήδη υπάρχει η πολιτική συμφωνία. Η Προεδρία θα ασκήσει όθηση προς την κατεύθυνση αυτή. Τέλος, Μποργέζιο, Έχω εν μέρει απαντήσει στην ερώτησή σας για προληπτικά μέτρα. Διάλογος και πέραν των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή ε, ε, ανάμεσα στην μεταναστευτική πολιτική και την πολιτική αναπτύξεως. Στο Μάλμε θα συζητήσουμε σχετικά στο ε, Συμβούλιο Υπουργών εκεί. Με, θα προσκαλέσουμε βέβαια και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσης να συμμετάσχουν στο διάλογο αυτό. Σας ευχαριστώ για τις συγκεκριμένες αλλά και ταχύτατες κατά τα άλλα παρατηρήσεις σας. το θέμα της διαχείρισης του χρόνου είναι πολύ, ε, θα έλεγα, σημαντικό. 1,5 λεπτό το πολύ 2 λεπτά γιατί έχουν ζητήσει 20 μέλη τον λόγο και δεν προλάβουμε. Σας θυμίζω λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να είσαστε συνοπτικοί. να ξεκινήσω λέγοντας ότι λέει η κυρία Κοράτσα Μπίλτ που βλέπω τον κύριο Μπίλστρομ εδώ. Ο κύριος Μπίλστρομ είναι πραγματικά ικανότατος στο να διαχειριστεί θέματα ανθρωπιστικά, θέματα αλληλεγγύης αλλά και θέματα παράνομων συμπεριφορών και καταστάσεων. Συνδυασμός δηλαδή δύο πραγμάτων που πρέπει να να προωθήσουμε και εδώ στην Ευρώπη. Το σουηδικό παράδειγμα νομίζω ε, είναι αρκετά καλό. Έχει βοηθήσει ε, και στην ένταξη των μεταναστών ε, στη χώρα μου. Τώρα για την εκπαίδευση των υπευθύνων υπαλλήλων που ασχολούνται με τα του ασύλου. Θα θέλατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες περισσότερες για το πού βρίσκεται η συζήτηση στο Συμβούλιο. Εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Επιτροπή μας να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που, ε, θέσατε το θέμα της απελευθέρωσης των θεωρήσεων για τα Δυτικά Βαλκάνια και για το χρονοδιάγραμμα το οποίο προτείνεται. Είπατε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα υιοθετηθούν νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και ελπίζω το Κοινοβούλιο να μην καθυστερήσει γραφειοκρατικά και συνεχίζουν εκατοντάδες χιλιάδες Ευρωπαίοι να νιώθουν φυλακισμένοι στις χώρες τους. Ελπίζω ότι η Επιτροπή μας θα μπορέσει να καταλήξει πριν το τέλος του χρόνου. Κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μας ρωτούν συχνά οι πολίτες και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη ερώτηση ε, στην πραγματικότητα, με τρόπο να απαντήσουμε δηλαδή με άλλη ερώτηση. Στην πραγματικότητα πρέπει να ρωτήσουμε τι κάνουν οι κυβερνήσεις και τι κάνουν οι υπουργοί, οι εθνικοί υπουργοί. Αυτά που είπε ο κύριος ε, υπουργό δεν αποτελούν πάντοτε εγγύηση για το γεγονός ότι οι υπουργοί που εγκρίνουν την κοινή θέση του Συμβουλίου την εφαρμόζουν κιόλα στις πατρίδες τους. Πρόκειται για μια εμπειρία την οποία κάνουμε σε πολλές χώρες μέλη. Ότι δηλαδή η εφαρμογή της ε, κοινή θέσης στην πραγματικότητα χωλαίνει στις ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγμα του κυρίου Μπερλουσκόνη που συμφωνεί αλλά όταν πρόκειται για επαναπροώθηση προσφύγων στην Λιβύη κάνει άλλα πράγματα. δεν τηρεί τα συμφωνηθέντα, δεν τηρεί τις διαδικασίες. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι αφενός ποιες δυνατότητες έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσουμε ορισμένες νομικές διαδικασίες. Και σε ό,τι αφορά την παράνομη μετανάστευση, εγώ έχω μια άλλη ερώτηση. Δηλαδή, πόση πεποίθηση έχει η Σουηδική Προεδρία ότι θα καταλήξει πραγματικά σε δεσμευτικές ποσοστώσεις ώστε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι υποχρεωμένοι να διαφύγουν από τις χώρες τους διότι διώχονται, θα γίνουν ε, δεκτοί στις χώρες μέλη. Και βεβαίως πρέπει να ελαφρυνθεί το βάρος το οποίο φέρουν οι νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς και πρέπει να μοιραστούν οι πρόσφυγες σε όλες τις χώρες. Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολικό το βάρος αυτό για τις υπόλοιπες Νομίζω ότι μια δίκαιη κατανομή δεν θα επιβαρύνει τις χώρες. Εκτός τούτου είμαι πεπισμένη ότι με μια τέτοια δίκαιη κατανομή θα μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθάρι στο οικοδόμημα της ε, καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης. Διότι η παράνομη μετανάστευση είναι και απαράδεκτη, αλλά και όταν γίνεται σε μεγάλους αριθμούς υπονομεύει και την διάθεση των ε, λαών να υποδεχθούν και νόμιμους μετανάστες. Λουί Μισελ. Θα πρέπει να κάνουμε μια ξεκάθαρη διάκριση εδώ ανάμεσα στην προβληματική της μετανάστευσης και αυτήν του ασύλου η μία έννοια θα έλεγα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εξυπηρετεί με πλάγιο τρόπο την άλλη. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα έλεγα με κάνει να ανησυχώ λίγο, για το οποίο δεν άκουσα πολλά πράγματα. Δεν άκουσα τίποτα. Κύριε Υπουργέ, φάνηκε ότι ανησυχείτε ιδιαίτερα για να καλύψετε τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό των ευρωπαϊκών χωρών και καταλόγω, κατανοώ την στάση αυτή, αλλά δεν άκουσα τίποτα για το θέμα και την προβληματική της φυγής των εγκεφάλων. Οι χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες έχουν πάρα πολλά προβλήματα με το λεγόμενο brain drain και αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα. γιατί στην ουσία εσείς θέλετε να εκενώσετε τις χώρες από την Αφρική, από την Ασία και τα λοιπά, από μηχανικούς, από γιατρούς, από νοσοκόμες. Και όμως εμείς με τη λογική μας, με το που βγαίνουν από τις σχολές τους, στην ουσία ε, τις κλέβουμε, τους κλέβουμε από τις χώρες τους. Και εγώ διαμαρτύρομαι για αυτή την διάσταση της πολιτικής μας. Αν θέλουμε πράγματι να σεβαστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το πρόβλημα, γιατί οι θέσεις σας είναι υπερβολικά πραγματιστικές και οι θέσεις σας είναι ηλιστικές θα έλεγα, ε, καλύπτοντας τα συμφέροντα αποκλειστικά των ε, χωρών των ευρωπαϊκών. Ίσως υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να ανταποκριθούμε στην έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού από το να αδειάζουμε, θα έλεγα, τις χώρες της υποανάπτυξη από τα στελέχη τους. Η κυρία Παπαδοπούλου. Κύριε Υπουργέ, έχετε κάνει σωστέ διαπιστώσει για τη Μεσόγειο και έχετε δώσει πολύ εύστοχες απαντήσει. Ρώτησα τη συνάδελφό σα, Υπουργό, προηγουμένω και δεν πήρα απάντηση. Έτσι επανέρχομαι με μια παρόμοια ερώτηση. Η Κύπρος είναι μια από τις χώρες της Μεσογείου που είναι άμεσα εκτεθειμένη σε πιέσεις λόγω παράνομης μετανάστευσης στις ελεύθερες περιοχές δεχόμαστε ένα αυξημένο αριθμό παράνομων μεταναστών και αιτητών ασύλου από τρίτες χώρες. Γιατί η στρατηγική θέση της χώρας μου είναι τέτοια που θεωρείται ως γέφυρα ανάμεσα στις τρίτες χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρόβλημα όμως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, θα έλεγα τραγικό, στις κατεχόμενες περιοχές. Γνωρίζετε ότι από το 1974 μέχρι σήμερα για 35 συναπτά έτη, υπάρχει κατοχικό στρατός, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να ασκήσει έλεγχο και να εφαρμόσει στα κατεχόμενα ευρωπαϊκά εδάφη το ευρωπαϊκό κεκτημένο και εκεί τα πράγματα είναι ανεξέλεκτα. Υπάρχει ακριβώς λάθρομετανάστευση που είναι εκτός ελέγχου και ταυτόχρονα παράνομος επικισμός από την Τουρκία προς τις κατεχόμενες περιοχές. Υπάρχει έξαρση της παραοικονομίας. Όλα αυτά τα καταγγέλλω. Για να εφαρμοστούν όσα έχετε πει, χρειάζεται πολιτική βούληση. Χρειάζεται η κατοχική Τουρκία να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία και να συνεργαστεί. Αυτό δεν υπάρχει. Και η Τουρκία δεν εφαρμόζει το πρωτόκολλο για να σεβαστεί ότι αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Επομένως, οι ερωτήσεις μου σε εσά είναι ξεκάθαρες. Η πρώτη είναι η εξής πρέπει η Τουρκία να μείνει στο απειρόβλητο μέχρι ότου βρεθεί η πολιτική λύση στο Κυπριακό, τι θα κάνει ο κύριος Μπαρό όταν θα επισκεφτεί σε λίγες μέρες την Τουρκία. Θα ασκήσει πιέσεις. Και η δεύτερη ερώτηση. Εφόσον η Τουρκία θέλει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έπρεπε να ασκηθούν πιέσεις ώστε να συμμορφωθεί, να σεβαστεί τις ευρωπαϊκές αξίες τις ευρωπαϊκές ανησυχίες και τις διεθνείς υποχρεώσεις και να αναγνωρίσει επίσημα την Κυπριακή Δημοκρατία ώστε να δράσουμε προληπτικά και να σταματήσει η παράνομη μετανάστευση. Αναμένω τις εύστοχες και σύντομες απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Mrs. Head, please. Tack så mycket ordförande och tack minister Billström för din intressanta presentation. Jag önskar dig riktigt lycka till med det svenska θα ήθελα και εγώ να σας απευθύνω τις θερμότερες ευχές μου για επιτυχίες στην προσπάθειά σας. Τα θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα θα έχουμε ελπίζω τη δυνατότητα να τα ξανασυζητήσουμε. Να προσθέσω ένα επιμέρους θέμα, το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών. Το θέμα των δικαιωμάτων των παιδιών θα πρέπει να γίνει πιο σημαντικό, ιδιαίτερα μετά την υιοθέτηση της συνθήκης της Λισαβόνας ένα σοβαρότατο πρόβλημα είναι το θέμα των παιδιών μεταναστών που έρχονται μόνα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα και πώς θα το αντιμετωπίσετε στο μέλλον. Σχετικά με το θέμα της επιστροφής των προσφύγων αυτών, της επαναπροώθησης κτλ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επανεξετάσουμε για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται Grazie per la relazione che ci ha fornito oggi il Ministro. Η κυρία Σερακιάνη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσίαση την οποία μας κάνει σήμερα. Ξέρετε ότι χθε ο Πρωθυπουργό της Ιταλίας είπε ότι θα μπλοκάρει τις εργασίες του Συμβουλίου αν εξακολουθήσουν οι εκπρόσωποι τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες να σχολιάζουν τον τρόπο αντιμετώπισης των παράνομων μεταναστών με τον τρόπο που το κάνουν μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι σκοπεύετε να κάνετε, ιδιαίτερα μετά από τα σχόλια τα οποία έκανε ο κύριος Μπαρό για αυτούς που έρχονται από τη Λιβύη. Ευχαριστώ η κυρία Μπλανκεβιτσίουτε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσία των προτεραιοτήτων της Σουηδικής Προεδρίας. Να μου επιτρέψετε να θέσω ορισμένες ερωτήσεις. Οι 130 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζήτησαν από την Ένωση να αποκτήσουν ε, περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της μετανάστευσης. Οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση το πρόβλημα επιβεβαιώνουν ότι η νόμιμη μετανάστευση είναι ευεργετική για την επίλυση πολλών προβλημάτων αλλά ε, οι αρνητικές επιπτώσεις από την παράνομη μετανάστευση γίνονται αισθητέ στις μεγάλες αστικές συγκεντρώσεις και γι' αυτό ακριβώς οι εκπρόσωποι των μεγάλων πόλεων ζητούν περισσότερες αρμοδιότητες για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτή θα ήταν μια πολύ καλή απάντηση και στα πλαίσια του προγράμματος της Στοκόλμης. Ξέρω ότι σε πάρα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις για απόκτηση περισσότερων εξουσιών από τις τοπικές αρχές στα θέματα της μετανάστευσης. Θα ήθελα όμως να μου πείτε την δική σας γνώμη. Το επόμενο θέμα έχει σχέση με τους μετανάστες οι οποίοι έρχονται να καλύψουν κενά στην αγορά εργασίας. σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλπάζει η ανεργία και αυτό δημιουργεί μερικές φορές κάποια προβλήματα. Είναι προφανές βέβαια ότι τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της υποδοχής των μεταναστών με ένα λογικό τρόπο και να προσαρμόσουν ακριβώς τις αφήξεις των μεταναστών στις ανάγκες της αγοράς εργασίας τους. Ε, υπάρχει και το θέμα του brain drain, δηλαδή της φυγής των εγκεφάλων από τις φτωχές χώρες και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ένα επιπλέον πρόβλημα είναι ότι πολλοί μετανάστες χρησιμοποιούνται από την εργοδοσία σαν φτηνό εργατικό δυναμικό και έτσι δημιουργούνται πολλά προβλήματα ανεργίας. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τις συγκεκριμένες μέχρι τώρα απαντήσεις τις οποίες δώσατε. Συγχαρητήρια. Ο κύριος Διάστε Μέρο. Αναγνωρίζω την σοφία της Επιτροπής αυτής στον τομέα της μετανάστευσης είναι προφανές ότι η φύση της παράνομης μετανάστευσης είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, όπως περίπλοκο είναι και το θέμα της αλλαγής της οδηγίας για το άσυλο. Πολλά από αυτά τα οποία είπατε βέβαια με βρίσκουν σύμφωνο. Έχω όμως ορισμένες, εξακολουθώ να έχω ορισμένες ανησυχίες. Ξέρετε ότι το πρόγραμμα της Χάγης θέτει το πρόβλημα της ε, ενσωμάτωσης, της ένταξης ε, και κάποια μέτρα τα οποία προτείνει πρέπει να τεθούν σε ισχύ από το 2010. Εσείς λέτε τώρα για το 2012. Πού είναι το πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα κοινή μεθοδολογίας, υπάρχει ένα πρόβλημα κατανομής του βάρους. Τι ακριβώς συμβαίνει ή μήπως υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες στο Συμβούλιο γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα του Ευρωπαϊκού Ταμείου ε, για τους ε, πρόσφυγες. Ε, πάρα πολύ λίγα χρήματα έχουμε στη διάθεσή μας και δεν προβλέπονται περισσότερα στα πλαίσια των δημοσιονομικών προοπτικών. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Υποτίθεται ότι με τα χρήματα αυτά θα ανοίξουμε και τα λεγόμενα γραφεία στήριξης των ετούντων άσυλο κτλ. Εμείς θα πρέπει να προωθήσουμε και να βελτιώσουμε τα μέτρα υποδοχής, όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά και για τους εκτοπισμένους κτλ. Περιμένω λοιπόν κάποιες περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη στάση της Σουηδικής Προεδρίας. Ε, ελπίζω να υπάρξει επιτέλους μια δημοσιονομική ενίσχυση του συγκεκριμένου αυτού ταμείου. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ο κύριος Μπόντες. Τα θέματα τα οποία συζητάμε σήμερα μου δημιουργούν θα έλεγα μια κάποια δυσθυμία. Να σας εξηγήσω γιατί πολλές χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης υφίστανται μια συντριπτική μεταναστευτική πίεση και παράλληλα δημιουργούνται συγκεντρώσεις των μεταναστών σε συγκεκριμένες περιοχές, ε, κάτι το οποίο επιτείνει τα προβλήματα αυτά. Λέτε ότι η μετανάστευση ανοίγει νέες ευκαιρίες και για τις ευρωπαϊκές οικονομίες μας. Μα τώρα αυτά δεν είναι έτσι. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, περιοχές μέσα στις Βρυξέλλες όπου είναι εντελώς κλειστές για τους Βέλγους, για τους κάτοικους της πόλης, τους πραγματικούς. Είναι μεταναστευτικά χωριά ουσιαστικά. Το ίδιο ισχύει και για τμήματα πόλεων όπως το Μάλμοε στην Σουηδία κτλ. Και όσο για τη φυγή των εγκεφάλων νομίζω ότι δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το θέμα είναι οι αριθμοί. Μπορεί να φτάσουν τα 50 εκατομμύρια οι παράνομοι μετανάστες που θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ανόητο και παράλογο να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να ενσωματώσει τέτοιου είδους υψηλούς αριθμούς. Το θέμα της απασχόλησης είναι σαφές. Ε, για να είστε 45 χρονών στην Ολλανδία και να βρεθείτε χωρίς δουλειά, τι δυνατότητες έχετε για να βρείτε δουλειά. Λοιπόν, Συν της άλλης επαναλαμβάνω ότι αυτές οι, οι απομονωμένες αστικές περιοχές τις οποίες κατοικούν οι μετανάστες είναι περιοχές τις οποίες το πολιτικό Ισλάμ, το φανατικό Ισλάμ βγάζει ρίζες και δημιουργεί επιπλέον προβλήματα. Έχω δύο επιπλέον ερωτήσεις λοιπόν. Συνειδητοποιείτε τα σοβαρά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν χώρες στο Παρίσι, όπως, ε, πόλεις όπως το Παρίσι, το Λονδίνο κτλ το Ρότερνταμ και είσαστε ε, προετοιμασμένος να αναθεωρήσετε τις πολιτικές σας σχετικά με τη δυνατότητα αυτών των 50 δίθεν εκατομμυρίων ε, που υποτίθεται θα βοηθήσουν τους κατοίκους της ε, Βορείου Αφρικής. Η κυρία Αντζελίλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την παρουσίαση του προγράμματος Υπάρχει μια πρόταση, όπως είναι γνωστό, για τη δημιουργία ενός προγράμματος ένταξης των προσφύγων. Είναι πολύ πιο συγκεκριμένο το θέμα έτσι όπως το θέτω, αλλά νομίζω ότι το πρόγραμμα αυτό καλό είναι σε επίπεδο σχεδιασμού, έχει μείνει όμως πάρα πολύ πίσω σε επίπεδο πραγμάτωσης. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να μένουμε τόσο πίσω, δεν θα πρέπει να καθυστερούμε τόσο πολύ, θα πρέπει να αποδείξουμε την πραγματική ιδέα που έχουμε στην Ευρώπη για την αλληλεγγύη και φυσικά η κατανομή του βάρους θα πρέπει να γίνεται με πιο δίκαιο τρόπο γιατί αλλιώς δεν είμαστε σε θέση να καλύψουμε τις ανάγκες των χωρών. Ιδιαίτερα λόγω του υψηλού αριθμού σε αυτή τη φάση των ετούντων άσυλο. Νομίζω λοιπόν ότι οι ευθύνε είναι πάρα πολύ ε, μεγάλες όλων των χωρών και δεν θα πρέπει οι περιφερειακές χώρες της Ένωσης όπως η Ελλάδα, η Ιταλία, η Μάλτα να υποφέρουν μόνες τους από τη μεταναστευτική πίεση. Όταν βλέπουμε να υπάρχουν μάλιστα συγκρούσεις μεταξύ χωρών όπως η Ιταλία και η Μάλτα, συγκρούσεις εννοώ διαφωνίες έντονες, και όταν βλέπουμε την τρομερή δυσκολία η οποία υπάρχει για το πού θα πρέπει να οδηγούνται τα σκάφη με παράνομους μετανάστες, το πρόβλημα δεν είναι θεωρητικό, είναι ένα πρόβλημα το οποίο επαληθεύεται σε καθημερινή βάση, μια τραγωδία που επαναλαμβάνεται καθημερινά. Το θέμα λοιπόν της υποδοχής των μεταναστών δεν θα πρέπει να το αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι χώρες οι περιφερειακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μεθοριακές, γιατί είναι σαφές ότι θα είναι ανάγκη ότι υπάρχει ανάγκη να κατανεμηθούν αυτοί που ζητούν άσυλο δίκαια και ισότιμα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουσα πολλά αρνητικά στοιχεία για τον τρόπο συμπεριφοράς των Ιταλών ή των Μαλτέζων, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι από τις ίδιες πηγές δεν έχω ακούσει τίποτα για τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες αγνοούν πλήρως το πρόβλημα και λέγουν πάρα πολύ απλά ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να υποδεχθούν ε, πρόσφυγες. Γι' αυτό λοιπόν όταν μιλάμε για ανθρώπινες ζωές τέτοιες συμπεριφορές είναι επικίνδυνες και απαράδεκτες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Αλφάνο. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό. Νομίζω ότι η κυρία Παπαδοπούλου έθεσε κάποιες ερωτήσεις και σήμερα το πρωί στις οποίες θα ήθελα να μας δώσετε πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Υπάρχει θα έλεγα μια έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν στη συγκεκριμένη περίπτωση και ε, η σύγχυση η οποία δημιουργείται δεν είναι πάρα πολύ, ε, ε, πάρα πολύ χρήσιμη στη συγκεκριμένη φάση. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι μια Ιταλική εφημερίδα έγραψε πρόσφατα, έδειξε μάλλον κάποιες πάρα πολύ ενοχλητικές φωτογραφίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι Σομαλοί πρόσφυγες στο στρατόπεδο Γκαντούφα της Λιβύης. Αυτοί ήταν Σομαλοί οι οποίοι συνελήφθησαν μόνο και μόνο γιατί προετοίμαζαν την μετάβασή τους στο Ιταλικό νησί Λαμπεντούζα. και αντιμετωπίστηκαν σαν εγκληματίες ουσιαστικά, σαν κακοποιοί, με ό,τι συνέπειες έχει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, η κατάσταση στη Λιβύη είναι φρικτή για τους ανθρώπους αυτούς. 60 πρόσφυγες στριμώχνονται σε ένα κελί. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες και επαναπροωθούνται στη Σομαλία πολλοί από αυτούς με απόλυτα βίαιο και απάνθρωπο τρόπο. και γι' αυτό ε, κάποιοι από αυτούς μάλιστα δεν θα έπρεπε να επαναπροωθηθούν γιατί είχαν ήδη ζητήσει ε, πολιτικό άσυλο. Αλλά δυστυχώς η πλευρά της Λιβύης δεν τα καταλαβαίνει αυτά, συμπεριφέρεται με απαράδεκτο τρόπο Και εγώ μάλιστα σήμερα το απόγευμα πριν έρθω εδώ άκουσα από τον εκπρόσωπο της Διεθνούς Αρμοστίας για τους πρόσφυγες ότι δεν μπόρεσε να επισκεφτεί η Διεθνής Αρμοστία τους πρόσφυγες στην χώρα αυτή. Πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πολύ σοβαρά εάν η πολιτική της Ιταλίας στα θέματα της μετανάστευσης είναι συμβατή με την κοινοτική πολιτική ο τρόπος με τον οποίο επιτελείται η επαναπροώθηση των παρανόμων αυτών μεταναστών είναι συμβατός με τα διεθνώς ισχύοντα. Πρέπει να μας δώσετε μία απάντηση σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σαν εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλετε να πάτε στη Λιβύη, να προσπαθήσετε να πάτε στη Λιβύη για να δείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω όπως είπα και στην αρχή της παρουσίασής μου ότι τέθηκε η ερώτηση και από μένα το πρωί και από άλλους συναδέλφους, αλλά απάντηση δεν δόθηκε. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε μια απάντηση και δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την προτροπή του Μπερλουσκόνη και να μην λέμε κουβέντα. Σας παρακαλώ να σεβαστείτε το χρόνο από εδώ και πέρα. Κέλλερ. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι υπάρχει ανάγκη να προωθηθούν πρωτοβουλίε για την κοινή διαδικασία ασύλου, που δεν θα πρέπει όμως να κινηθεί στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Και επίση, πώς θα αντιδράσετε εάν οι χώρε μέλη δεν πληρούν την, ε, δεν σέβονται την συνθήκη της Γενέβης ή δεν εξασφαλίζουν δίκαιες διαδικασίες για αυτούς που ζητούν άσυλο. Και πώς θα αντιδράσετε αν οι αντιδράσεις δεν γίνουν αποδεκτές από τις χώρες μέλη που θίγονται. Το πρόγραμμα της Στοκόλμης προβλέπει πολλά σχετικά με την ε, συλλογή δεδομένων προσωπικών δεδομένων, ε, για παράδειγμα για δακτυλικά αποτυπώματα μεταναστών κλπ. Και η εξασφάλιση προσωπικών, της προστασίας προσωπικών δεδομένων των μεταναστών που ίσως να μην είναι πολίτες ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι πάντως ανθρώπινα όντα και έχουν και αυτά ανάγκη προστασίας. Μαστέλα. Ε, Πιστεύω κύριε Πρόεδρε ότι υπήρξε μια επίδειξη θα έλεγα πολιτικού θάρρους από πλευράς της Σουηδικής Προεδρίας σε σχέση με τις ε, δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικό το θέμα γιατί όλα αυτά άπτονται της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Η Ευρώπη φυσικά δεν έχει μία φωνή στον συγκεκριμένο τομέα. Είναι πολλές φορές κάποια προβλήματα τα οποία κυριαρχούν, τα οποία έχουν αυστηρά οικιακό θα έλεγα εθνικό χαρακτήρα. Η τραγωδία η οποία εκτιλήσεται στις ακτές της Μάλτας και της Ιταλίας δεν μπορεί παρά να αφορά και την υπόλοιπη Ευρώπη και το Βερολίνο. Και μέχρι τώρα η ευρωπαϊκή δημοκρατία αγνοεί το πρόβλημα. Και μάλιστα όχι μόνο το αγνοεί, αλλά ακούγονται πολλές φορές μεγάλα λόγια και υποτίθεται ότι θα βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι φτάνουν στην Ευρώπη, αλλά δυστυχώς τα λόγια αυτά δεν εξυπηρετούν κανένα. Και ακούγονται μόνο οι φωνές της Ευρώπης από τους εκπροσώπους τύπου. Οι εκπρόσωποι τύπου πρέπει να μιλάνε, δεν διαφωνώ εγώ με αυτό. Και νομίζω ότι η γραμμή την οποία ακολουθεί η Ιταλική κυβέρνηση είναι μια γραμμή η οποία ναι δεν έχει συζητηθεί αλλά δεν θα πρέπει να στρέφουμε την προσοχή μας μόνο στη στάση των Ιταλών και της Ιταλικής κυβέρνησης και να αγνοούμε ε, το δράμα το οποίο επαναλαμβάνω εκτιλήσεται στη Μεσόγειο. Ίσως θα πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία η Σουηδική κυβέρνηση σε συνεργασία με τις χώρες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, το βασικό πρόβλημα, έτσι ώστε ο καθένας να μην αντιμετωπίζει το πρόβλημα μεμονωμένα, να μην παραβιάζει την γραμμή την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει και τότε θα υπάρξει λιγότερο δράμα για τις φτωχές αυτές ψυχές οι οποίες πολλές φορές χάνουν τη ζωή τους προσπαθώντας να έρθουν στην Ένωση. Λοιπόν, σας θυμίζω να διαχειριστείτε το χρόνο καλύτερα. Ο κύριος Μπρόνς. Πάρα πολλοί πρόσφυγες γενικότερα προσπαθούν να ξεφύγουν από καταστάσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Αλλά πολλές φορές όταν έρχονται στις χώρες υποδοχής πάβουν να είναι πραγματικοί πρόσφυγες και μετατρέπονται σε απλούς οικονομικούς μετανάστες. Νομίζω ότι είναι απόλυτα φυσικό κάποιες χώρες να ακολουθούν μία μορφή θα έλεγα αυτόνομης πολιτικής. Ξέρετε ότι η σωματεμπορία σαν παράδειγμα έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία α, εν πολλής επηρεάζουν και προσωμιάζουν προς τις μεταναστευτικές ροές. Τι εννοώ με αυτό. Υπάρχει η παγκοσμιοποίηση που επιβάλλει ορισμένους κανόνες και οι μετανάστες αντιμετωπίζονται όχι σαν ανθρώπινα όντα, αλλά σαν απλά στοιχεία της παραγωγής. Χωρίς μικρόφωνο, επόμενος ομιλητής. μία ερώτηση που βασίζεται σε μία δευτερεύουσα παρατήρηση που κάνατε πριν ότι το ΣΥΣ 2 δεν είναι ακόμα λειτουργικό. Γιατί όχι παρόλες τις καθυστερήσεις και τι έχει σκοπό να πράξει η ε, Προεδρία ώστε να καταστεί λειτουργικό. Και τρίτο, μετά από την μακρά αυτή καθυστέρηση, πότε θεωρείτε ότι θα μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Θα αρχίσω με την κυρία Κορατσαμπίλ, την οποία ήθελα να ευχαριστήσω για τα ευγενικά της λόγια. Όσον αφορά το Γραφείο Υποστήριξης και την θέση του Συμβουλίου, μετά την άτυπη συνάντηση του Ιουλίου, πιστεύω ότι όλα τα κράτη-μέλη συμφώνησαν να δημιουργηθεί αυτό το γραφείο υποστήριξης. Είναι σαφής η θέση του Συμβουλίου. Και ξεκινώντας από αυτή τη βάση μπορούμε να συνεχίσουμε τις συζητήσεις του Κοινοβούλιο. Το θέμα των θεωρήσεων επίσης είναι πολύ σημαντικό. Σα είπα ότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία δεν συμφωνούν με τα μέρη ελέγχου τα οποία έχουν οριστεί στο χάρτη μέχρι τώρα σχέση με αυτό το οποίο είπε τώρα η κυρία Κέλλερ, δηλαδή πώς μπορούμε να φτάσουμε σε ένα, στη δημιουργία ενός κοινού συστήματος ασύλου, επιμένω, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα εκπονηθεί και θα παρουσιαστεί η οδηγία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει κάποιες προϋποθέσεις και θα μπορούσε ενδεχομένως να υπάρξει και ένα, ένας διάβλος συνεργασίας στα πλαίσια της χορήγησης ασύλου μεταξύ των κρατών, η ίδια η Κομισιό είναι εκείνη η οποία πρέπει να θέσει το γενικότερο πρέσιο. Η Κομισιό και τα αρμόδια. Τώρα, μεταξύ των κρατών μελών, σίγουρα πρέπει να γίνει καλύτερη κατανομή των ετούντων άσυλο. Μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να καθορίσουμε τις βέλτιστες συνθήκες για να γίνει κάτι τέτοιο, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν κάποια σχέδια για να δούμε στη Μάλτα Φερρυπίν πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα λόγω της θέσης της ο κύριος ε, Μισελ έφυγε. Θα ήθελα όμως ε, να απαντήσω στο ερώτημά του. Το θέμα αυτά που er, το θέμα αυτό το οποίο έφυξε θα ήθελα να αναφέρω για την φυγή εγκεφάλων και σε κοινοτικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να αντισταθμίσουμε τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται λόγω ελλείψεων που έχουμε ε, σε έργα υποδομής στον τομέα της υγείας, Και πολλές φορές πρέπει να πω ότι σε κάποιες χώρες επικρατούν κάποιες απόψεις τις οποίες ακόμη θα μπορούσα να πω ότι είναι απικιακού τύπου. Το να σκεφτεί κανείς ότι δεν μπορεί μία νοσοκόμα από την Τανζανία να πάει να δουλέψει κάπου αλλού είναι πολύ πατριαρχικό ως σκεπτικό. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε τέτοιου είδους νοοτροπίες. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι τα εμβάσματα των μεταναστών στις χώρες του. Πράγμα που βοηθά τις χώρες και αυτές κάπως οικονομικά να αναπνεύσουν. Αυτό μπορούμε να το αρνηθούμε. Και αυτό είναι ένα από τα καλά της ε, μετανάστευσης. Σήμερα υπάρχει πρόβλημα με την κρίση και με την αγορά εργασίας παντού. Αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το πρόβλημα το δημογραφικό. Κυρία Παπαδοπούλου, εσείς αναφέρατε τα προβλήματα της Κύπρου. Το συνειδητοποιούμε ότι έχετε πρόβλημα και θέλουμε να ευρεθεί ολική λύση, συνολική λύση στο πρόβλημα της Κύπρου. Ή ούτως ή άλλως να βελτιωθεί η παρούσα κατάσταση, αν δεν μπορέσει να ευρεθεί ολική λύση. Όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή το κείμενο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών, το οποίο υπάρχει στην θεωρία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτό το τομέα και με την επόμενη Προεδρία, με την Ισπανική, θα προετοιμάσουμε κάτι για αυτό το θέμα και στα πλαίσια του προγράμματος Στοκχόλμης δεν θα τα ξεχάσουμε τα παιδιά. Τώρα, όσον αφορά το οποία είπε η κυρία Σερακιάνη. Δεν μπορώ ίσως να προφέρω ε, πολύ καλά τα ονόματά σας. Σε σχέση με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπερλουσκόνη, η Επιτροπή προσπαθεί να λάβει υπόψη τις αρχές και τους κανόνες που περιέχονται στην οδηγία. Στην κυρία Βατροβιτσούτε θα πω ότι όντως θα πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταβάλλεται και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές. Προσπάθησα στις απαντήσεις που σας δίνω να εξηγήσω πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα αγορά εργασίας οι μετανάστες για δουλειές τις οποίες δεν θέλει να κάνει κανένας από εμάς. Αλλά θα πρέπει να εργάζονται χωρίς να την χάνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης. Κύριε Δίαθ Δεμέρα, στα πλαίσια του προγραμμάτου της Χάγης και την προσωρινή υποδοχή, θα πω το εξής. Πέρσι το Δεκέμβριο οι ε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είπαν ότι θα πρέπει να υπάρχει μία προθεσμία για την ε, ε, δημιουργία αυτού του γραφείου υποστήριξης. Με ημερομηνίες 2010-2012. Πότε είπατε θα αρχίσει να λειτουργεί αυτό το κέντρο υποστήριξης. Ελπίζουμε ότι τα πραγματικά μέτρα υποστήριξη τη μετανάστευση θα μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή από το 2012 και μετά. Επίσης πρέπει να πω ότι υπάρχουν πολλά εκατομμύρια δυνητικών εργαζομένων παντού που περιμένουν δουλειά. Η Σουηδία σε αυτή την περίοδο της κρίσης πρέπει να σας πω ότι χρειάζεται εργατικά χέρια σε κάποιους τομείς, παρά την κρίση. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες, αλλά στην δική μας ακόμη χρειαζόμαστε τους μετανάστες. Και βεβαίως είναι πρόκληση η υποδοχή των μεταναστών, αλλά για κάποιες δουλειές χρειαζόμαστε τους μετανάστες. Θα πρέπει λοιπόν τα συστήματα υποδοχής των μεταναστών να βασίζονται στις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξετάσει κάθε χώρα χωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες της, για να μπορέσει να βρει λύσεις. κυρία Αλφάνο, ε, θα πω το εξής. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν σαφείς κανόνες, το επαναλαμβάνω, και να γίνονται σεβαστές οι αρχές του ασύλου από όλους και για όλους. Και βεβαίω θα πρέπει να ισχύει η αρχή της αμοιβέ και της δίκαια συνδρομή. Υπάρχουν άτομα στα οποία δεν έγινε αποδεκτή η αίτηση ασύλου. Και βεβαίως και από την ε, Λιβύη θα πρέπει να ζητήσουμε να κάνει σεβαστούς τους κανόνες. Θα πρέπει λοιπόν μέσω της ε, ε αντιπροσωπείας μας στη Λιβύη να στείλουμε κάποια σαφή μηνύματα στη χώρα αυτή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι απάντησα σε περισσότερα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν. Σχεδόν σε όλα απάντησα. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ μίλησα και για τα θέματα της δικής μου αρμοδιότητας, αν αναφέρθηκε και στις θέματα αρμοδιότητας της συναδέλφου Μπέτρη Σάσκ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονό ότι σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι έλαβαν το λόγο και έκαναν ερωτήσεις, θα θέλαμε τελειώντας να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό για τις λεπτομεριακέ απαντήσεις που έδωσε. Κύριε Υπουργέ, προσβλέπουμε σε περαιτέρω συνεργασία μαζί σας κατά τη διάρκεια της Σουηδική προεδρία και σας χαιρετούμε ευχόμενοι και καλή τύχη.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 Eurojust. Okay, you will give the floor to López Mañana, mañana, por la tarde. Call eight No, the, the previous, the previous. Eh, Libre. Teresa.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 Θα uh, συμφωνήσετε μαζί μου ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρέπει να βιαστούμε λοιπόν. Ας περάσουμε στο επόμενο θέμα, την παρουσίαση δηλαδή από τον πρόεδρο του Eurojust, τον κύριο Χωσέ Λουίς Λόπες Ταμότα, ο κύριος Μπουσουτήλη ζητάει το λόγο. Αν κατάλαβα καλά, σήμερα το πρωί συμφωνήσαμε ότι αμέσως μετά την παρουσίαση του Σουηδού Υπουργού θα συζητούσαμε το θέμα της γνωμοδότησης για τον προϋπολογισμό. Έχει υπάρξει μια αλλαγή. Δεν ξέρω, αν θυμάμαι καλά, εγώ ο ίδιος είχα προτείνει την αναβολή του θέματος αυτού για να γίνει μετά το Eurojust. Έτσι ώστε να είναι όλα τα μέλη παρόντα και να είναι σε θέση να υποβάλουν τις προτάσεις τους για την πρόταση γνωμοδότησης για το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Αν δεν σας πειράζει λοιπόν, αμέσως μετά την παρουσίαση του κυρίου Νταμότα θα μπορέσουμε να αφιερώσουμε μισή ώρα να ακούσουμε τον κύριο Λόπες Ταμότα. Επαναλαμβάνω ότι το Eurojust είναι ένα όργανο με πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Ε, σαφές είναι ότι στρέφουμε την προσοχή μας στις επιδόσεις αυτού του οργάνου και η παρουσία του Προέδρου του Eurojust είναι πλέον παραδοσιακή θα έλεγα στην Επιτροπή μας τα τελευταία χρόνια. Περιμένουμε λοιπόν εμείς να ακούσουμε για έβδομη φορά τον Πρόεδρο του Eurojust, τον κύριο Χωσέ Λουίς Νταμότα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αγαπητά μέλη, είναι μεγάλη τιμή για μένα και μεγάλη χαρά που με προσκαλέσατε και είμαι παρόν στη συνάντησή σας σήμερα για να παρουσιάσω την έκθεση για τις δραστηριότητες της Eurojust προς τα νεοεκλεγέντα μέλη της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών. Εκ μέρους του Eurojust θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λόμπες Αγγιλάρ, για την εκλογή σας στην Προεδρία. Λέγομαι Ζωζέ Λόπες Νταμότα, είμαι Πορτογάλος, μέλος της Eurojust, είμαι βοηθός Γενικού Εισαγγελέα στην Πορτογαλία και έχω εκλεγεί πρόεδρος του Eurojust τον Νοέμβριο του 2007. Ακριβώς με την ιδιότητα αυτή είμαι μπροστά σας σήμερα για να σας παρουσιάσω την 7η ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων του Eurojust. Όλοι σας έχετε αντίγραφα της έκθεσης της γλώσσας, σας, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θα παρουσιάσω την έκθεση αυτή λεπτόμερος, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχει γραπτά θα ήθελα όμως να χρησιμοποιήσω τον χρόνο τον οποίο έχω στη διάθεσή μου να, για να σας ενημερώσω για τις παρούσες δραστηριότητες της Eurojust το 2008 και το 2009 και για τις εξωτερικές σχέσεις του Eurojust, ένα σημαντικό τομέα, και να αναφερθώ και στο μέλλον του Eurojust στα πλαίσια των νέων αποφάσεων που κυκλοφόρησαν στις 4 Ιουνίου του 2009. Αυτή η νέα απόφαση θα καταστήσει το Eurojust αποτελεσματικότερο και θα επανέλθω αργότερα στην παρουσίασή μου στα θέματα αυτά. Ας μου επιτρέψτε μου λοιπόν να επαναλάβω τους τρεις βασικούς στόχους του Eurojust. Πρώτον, να καλύψουμε τις ε, <clears throat> δικαστικές αρμοδιότητες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ποινικό τομέα. Αυτό αποφασίστηκε ήδη από το 2002 σαν προσωρινό Eurojust. Υπήρξε ένα άλλο θέμα το οποίο είναι ο συντονισμός των αρμόδιων εθνικών αρχών και το τρίτο θέμα που είναι θα έλεγα και το raison d'être του Eurojust είναι να δώσουμε κίνητρα για καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στις εθνικές αρχές όταν έχουν να αντιμετωπίσουν διαμεθοριακές υποθέσεις που να περιπλέκουν, που να εμπλέκουν, συγγνώμη, καλύτερα άνω των δύο χωρών. Βασικός στόχος είναι να βελτιώσουμε την συνεργασία, εν πάση περιπτώσει, ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να βελτιώσουμε τις ανακριτικές και διοκτικές δραστηριότητες όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα όπως τη διεθνή δημοκρατία, τη σωματεμπορία, το εμπόριο ναρκωτικών και να πετύχουμε να φέρουμε γρήγορα και αποτελεσματικά τους εγκληματίες στη δικαιοσύνη. Δεν είμαστε ανακριτικό σώμα, δεν είμαστε δικαστικό σώμα, απλά ασχολούμεθα με θέματα δικαστικής συνεργασίας και ρόλος μας είναι να υποστηρίξουμε και να βοηθήσουμε τις προσπάθειες που κάνουν τα, ε, τα κράτη-μέλη. Για τις αρμοδιότητές μας 2008 και 2009, να μου επιτρέψετε να επιμείνω σε ορισμένα θέματα. Αν δείτε και τη γραπτή μας έκθεση, θα δείτε ότι ήδη από το 2002 το Eurojust έχει κάνει αρκετά βήματα πρόοδο για τα ναρκωτικά, για την καταστροφή περιουσίας, για τις απάτες. Είναι περιπτώσεις με τις οποίες έχουμε ασχοληθεί στο Eurojust. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι οποίες παραπέμπονται στο... ο αριθμός μάλλον των υποθέσεων που παραπέμπονται στο Eurojust αυξάνονται κατ' έτος. Το 2008 ασχοληθήκαμε με 1.819 υποθέσεις οι οποίες απεστάλησαν στο Eurojust από τα κράτη-μέλη. Αυτό αντιπροσωπεύει 10% αύξηση σε σχέση με το 2007. Ο αριθμός αυτός δεν είναι φυσικά ο μοναδικός δείκτης για τη συνεχιζόμενη επιτυχία του Eurojust. Γνωρίζουμε πολύ καλά, συνειδητοποιούμε πάρα πολύ ότι εξακολουθούμε να εργαζόμεθα σε ένα εντελώς ε, βασικό επίπεδο, απλό επίπεδο, ανταποκρινόμενοι σε αιτήσει αμοιβαία νομικής βοήθειας, συνδρομής. Πολλά μένει να γίνουν στις χώρες μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε όλες τις αποστολές και δράσεις του Eurojust όπως περιλαμβάνονται στις αποφάσεις οι οποίες έχουν ληφθεί για την ίδρυση του Eurojust του 2002. Η καταπολέμηση του διαμεθοριακού εγκλήματος απαιτεί σωστή συνεργασία. Όλοι συμφωνούν με αυτό. Αυτό υπάρχει και στο έγγραφα που τα ιδρυτικά, τα συστατικά του Eurojust αλλά αυτό είναι και το πιο δύσκολο πράγμα το οποίο μπορεί να πετύχει κανείς. Ο συντονισμός αυτός θα πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στις εθνικές αρχές διαφορετικών χωρών. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι μερικές φορές να υπάρξει αυτή η μορφή ε, ε, συνεργασίας και συντονισμού ανάμεσα στις ίδιες τις χώρες και στα διαφορετικά δικαστικά τμήματα, θα έλεγα, της ίδιας της χώρας ανάμεσα στους δικαστές, ανάμεσα στους ανακριτές και τους δικαστές, ανάμεσα στις εισαγγελίε και τους ανακριτές και τους δικαστές και πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε με υποθέσεις οι οποίες εμπλέκουν άνω των 10 μερικές φορές χωρών. Συνεπώς εδώ βρίσκεται και το κλειδί για μια σωστή συνεργασία ανάμεσα στις χώρες αυτές. Ο συντονισμός αυτός είναι απόλυτα απαραίτητος. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ελέγξουμε το επίπεδο των εγκληματικών δραστηριοτήτων που σοβούν στις χώρες μας. Θα πρέπει να καταπολεμούμε επίσης και αυτούς οι οποίοι εργάζονται προς το συμφέρον των εγκληματιών. Φυσικά θα διώξουμε κυρίως τα ίδια τα εγκληματικά δίκτυα. Αυτό το οποίο ελείπει όμως στην Ευρώπη, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή που αποτελείται από 27 χώρες και 23 γλώσσες, και 30 διαφορετικά νομικά συστήματα, αυτό είναι το πιο βασικό μας πρόβλημα, γιατί όταν ακριβώς έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση που εμπλέκει 10 ή 15 χώρες, έχουμε να αντιμετωπίσουμε 10 με 15 νομικά συστήματα και τα προβλήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μην αγνοήσω το πρόβλημα των οτροπιών και του νομικού πολιτισμού. Δεν θέλω τώρα εγώ να απαριθμίσω τις αρμοδιότητες του Eurojust, θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω την ιδέα του συντονισμού που περιλαμβάνεται στα ιδρυτικά άρθρα του Eurojust. Φιλοδοξία μας είναι να προχωρήσουμε στην αντιμετώπιση πιο περίπλοκων και δύσκολων υποθέσεων που να εμπλέκουν όσο περισσότερες γίνεται χώρες. Υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο θα ήθελα να υπογραμμίσω. την ανάγκη να δημιουργήσουμε δίκτυα δικαστικής συνεργασίας ήδη από το 2010 σε επίπεδο εισαγγελικό. Δεν είναι κάτι το οποίο οι ερευνητικές και προανακριτικές διαδικασίες δεν είναι μόνο, θα έλεγα, μονοπόλιο των διοκτικών αρχών, αλλά και των δικαστικών αρχών και των εισαγγελικών αρχών. Πρέπει να έχουμε περισσότερα μέσα στη διάθεσή μας για να είμαστε αποτελεσματικοί και να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των αστυνομικών αρχών, να παρεμβαίνουμε εκεί όπου είναι χρήσιμο και να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις ε, εγκληματικές οργανώσεις. Εδώ τίθεται και το θέμα του σεβασμού των αρχών, ή μάλλον των δικαιωμάτων των βασικών ε, των ε, προσώπων. Και εδώ απαιτείται έλεγχος των μέτρων τα οποία λαμβάνονται για το αν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και αυτό απαιτεί φυσικά καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές, στις αστυνομικές αρχές και στις δικαστικές αρχές. Αυτό είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό ενός κράτους δικαίου. Ε, μέχρι τώρα υπάρχουν ε, υποθέσεις στις οποίες η συμμετοχή μας σαν Eurojust ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Μπορώ να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Οδηγήσαμε στην διάλυση πολύ μεγάλων δικτύων ευρωπαϊκών σε μεγάλα δίκτυα παράνομης μετανάστευσης ε, στη διάλυση ενός πολύ μεγάλου δικτύου διανομής και εισαγωγής κοκαίνης κτλ. Οργανώσαμε πάρα πολλές ε, διαβουλεύσεις, επαφές ανάμεσα στις αστυνομικές αρχές και ε, προωθήσαμε τα θέματα της οργάνωσης ταυτόχρονων συλλήψεων σε διάφορες χώρες, όπως επίσης και δημεύσεων περιουσιών, ε, όλα αυτά είναι θέματα που πολλές φορές δύσκολα θα έλεγα εφαρμόζονται και ιδιαίτερα όταν πρέπει να γίνει ταυτόχρονα γιατί αν δεν γίνει κάτι τέτοιο μερικές φορές ταυτόχρονα τότε οι αποδείξεις ε, χάνονται. Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση έγιναν ταυτόχρονα 24 συλλήψεις σε πάρα πολλές χώρες. Σε μια άλλη περίπτωση συνελήφθησαν ταυτόχρονα 65, σε μια άλλη 42, και αυτά είναι τρία μόνο παραδείγματα. Το 2008 οργανώσαμε 132 συναντήσεις διαβούλευσης με την συμμετοχή των εθνικών αρχών, δηλαδή αστυνομικές αρχές, εισαγγελικές αρχές και δικαστές. Αυτοί είναι αυτοί που αποφασίζουν το τι πρέπει να γίνει και αυτοί συντονίζουν από ένα σημείο και μετά τη μορφή συνεργασίας τους. Σε αυτές τις συναντήσεις στις 132 του συντονισμού υπήρξε συμμετοχή άνω των 1500 εκπροσώπων των αστυνομιών, των δικαστικών σωμάτων και των εισαγγελιών. Αν δει κανεί τους αριθμούς των τελευταίων χρόνων λοιπόν θα καταλάβει ότι έχουμε οργανώσει σχεδόν 800 τέτοιες συναντήσεις συντονιστικές όπου έχουν εμπλακεί άνω των 6.000 εκπροσώπων αστυνομικών αρχών, δικαστικών αρχών και εισαγγελιών. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα σιγά σιγά σαν χιονοστιβάδα έχουν αρχίσει να γίνονται ορατά. Έχει μεγάλη σημασία να πούμε ότι το Eurojust θα πρέπει να ορίσει ακόμα καλύτερα τις λειτουργικές του ιδιότητες ε, υπό το φως των προτεραιοτήτων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ήδη από το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση εντοπίζει ορισμένες προτεραιότητες σε συγκεκριμένες μορφές εγκλημάτων και παρανόμων δραστηριοτήτων. Τομεί δηλαδή στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρέμβει με πλέον δραστήριο τρόπο. Δίκτυα δηλαδή πανευρωπαϊκά, σωματεμπορίας, έκπληνσης χρημάτων και απατών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο αλλά και τρομοκρατικών δραστηριοτήτων. Αυτό φαίνεται και στη δράση την εθνική της κάθε χώρας. Τα κράτη-μέλη συνειδητοποιούν τα ευεργετήματα θα έλεγα που μπορεί να προέλθουν από την συνεργασία αυτή Και εδώ μερικές φορές δημιουργείται ένα πρόβλημα γιατί οι προτεραιότητες αυτές πρέπει να είναι κοινέ και για τα κράτη-μέλη και για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν υπάρχει συντονισμός όμως σε όλες αυτές τις ενέργειες, κανένας δεν ελέγχει, κανένας δεν αξιολογεί, δεν αποφεύγονται επικαλύψεις και έτσι δαπανώνται, σπαταλώνται θα έλεγα οι πόροι τους οποίους έχουμε στη διάθεσή μας με παράλογο τρόπο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει εμείς να τεκμηριώνουμε καλύτερα τους τομείς τους οποίους παρεμβαίνουμε. Αν τυχόν μακρηγορώ κύριε Πρόεδρε να μου το υπενθυμίσετε, λίγο χρόνο ακόμα θέλω, υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις. Καταρχάς το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Το 2008 το Eurojust αντιμετώπισε 237 περιπτώσεις που εμπλέκουν την διευκόλυνση και τον συντονισμό διαδικασιών δικαστικών που οδήγησαν στην εφαρμογή του εντάλματος. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ο συγκεκριμένος κακοποιός ή ύποπτος μάλλον καταζητείται σε άνω των δύο ή τριών χωρών όπου θα πρέπει να αποφασιστεί ποια χώρα είναι αυτή η οποία θα προβεί στη σύλληψη. Το δεύτερο θέμα είναι η τρομοκρατία. Η τρομοκρατία είναι βασική προτεραιότητα, εξ αρχής ήταν βασική προτεραιότητα. Το Eurojust πάντα έχει προσπαθήσει να συνεισφέρει και στις προσπάθειες της Europol και νομίζω ότι είναι παραγωγική η στάση μας. Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το λεγόμενο Terrorist Convictions Monitor παρέχουμε αναλυτικές στατιστικές πληροφορίες ε, για τις τρομοκρατικές ιδέες οι οποίες υπάρχουν στην Ευρώπη. Φυσικά οργανώνουμε σε αιτήσια βάση και, συντον, και συναντήσεις των εθνικών συντονισμών για την, συντονιστών συγγνώμη, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Από το Σεπτέμβριο του 2005 και μετά υπάρχει μια καλύτερη θα έλεγα συνεργασία γιατί υποχρεώνονται οι χώρες μέλη να ενημερώνουν το Eurojust και έτσι συντονίζεται καλύτερα η, η κατάσταση, η οποία γενικότερα όμως παραμένει σε απαγοητευτικό επίπεδο, γιατί οι περισσότερες πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε είναι από ανοιχτές πηγές, δηλαδή πληροφορίες, τηλεόραση, πολύ περισσότερες πληροφορίες από ό,τι από τις εθνικές αρχές. Αυτό είναι η πραγματικότητα απογοητευτική. Οι ανακριτικές ε, θα έλεγα ενέργειες και διαδικασίες είναι απαραίτητες για την καταπολέμηση Φρουγετόρι. is not anymore ε, to fight the... Λοιπόν, αυτές οι μικτές ανακριτικές ομάδες είναι απαραίτητες για την βελτιωμένη αντιμετώπιση ε, του εγκλήματος. Έχουμε επίσης ε, και τη σύμβαση του Μαΐου του 2000 χρειάστηκαν πέντε χρόνια παρότι ελήφθη η απόφαση αυτή το 2000 για να εφαρμοστεί. Ήταν κάποτε ε, πραγματικά δύσκολο να θεωρήσει κανείς ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα τέτοιο μέσο, αλλά είναι τώρα πλέον ένα μέσο, ακριβώς αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση των μεικτών ανακριτικών ομάδων. Εδώ υπάρχει μια κάποια μορφή δυσθυμίας θα έλεγα γιατί υπάρχουν λίγες τέτοιες μικτές ανακριτικές ομάδες Έχουμε επίσης ε, χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξουμε με τη σειρά μας τις εθνικές αρχές για την δημιουργία ακριβώς αυτών των μεικτών ανακριτικών ομάδων, για να καλύψουμε τα έξοδα ταξιδίου των αστυνομικών, τα ξενοδοχεία τους, γιατί τα κράτη-μέλη λέει ότι δεν έχουμε χρήματα, λένε ότι δεν έχουμε χρήματα γι' αυτό, να τους δώσουμε διερμηνία, μετάφραση, υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Περιμένουμε τις αιτήσει των εθνικών αρχών. Είναι στην ιστοσελίδα του Eurojust και θα ήθελα να πω ότι έχει ήδη υπάρξει ένα σημαντικό αριθμό αιτήσεων, αλλά παρόλα αυτά η κατάσταση δεν είναι πάρα πολύ καλή. Ελπίζουμε οι τοπικές αρχές και η αστυνομία και οι δικαστές θα χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο μέσο καλύτερα για να καταπολεμήσουν το έγκλημα. Τέλος σχετικά με την, παιδική, με την προστασία της παιδικής ηλικίας. Ε, ε, το Συμβούλιο ζήτησε από την Eurojust να δημιουργήσει ένα σημείο επαφής, ένα contact point για την προστασία των παιδιών, για να μπορέσουμε να συντονίσουμε και να συλλέξουμε καλύτερα πληροφορίες από τις 27 χώρες και να δούμε ακριβώς ποια προβλήματα είναι αυτά τα οποία αφορούν τα παιδιά. Γνωρίζουμε φυσικά το πρόβλημα της παιδικής πορνογραφίας στο διαδίκτυο, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά και το κάνουμε αυτό σε αιτήσια βάση. αλλά τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας αυτής μέχρι τώρα δεν ήταν πιστικά. Ένα άλλο θέμα είναι οι εξωτερικές σχέσεις του Eurojust και αναφέρομαι εδώ τη συνεργασία είτε με άλλα ευρωπαϊκά σώματα είτε ε, με τρίτες χώρες. Προσπαθούμε να ορίσουμε με πρακτικό τρόπο τη συνεργασία μας με οργανισμούς όπως η Όλαφ, με υπηρεσίες μάλλον όπως η Όλαφ. Πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα για να είμαστε αποτελεσματικότεροι για την καπολέμηση της απάτης και άλλων μορφών τρομοκρατίας που άπτονται της προσβολής των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως την προστασία του Euro. Το Euro είναι ένα διεθνές νόμισμα και πρέπει να προστατευτεί από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα που να έχουν σχέση με την παραχάραξη των ευρώ. Και έχουμε επίσης και πάρα πολλά προβλήματα σχετικά με απάτες στα πλαίσια του κοινοτικού προϋπολογισμού. Εδώ υπάρχουν φυσικά και κάποιες παρανοήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες που έχει η Όλαφ από τη μία και το Eurojust από την άλλη. Λένε ότι το ίδιο είσαστε. Έτσι πιστεύουν πολλοί. Υπάρχουν όμως εδώ παρανοήσεις σχετικά με τον ρόλο των δύο οργάνων και θα πρέπει να ρυθμιστούν οι παρανοήσεις αυτές σχετικά τώρα με τη συνεργασία με το Europol. Είναι ο βασικός μας εταίρος, το Eurojust. Υπάρχει γιατί υπήρχε το Europol ή θα πρέπει να συνεργαστούμε φυσικά με την Ευρωπόλ, ε, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τη συμφωνία του 2004, να υπάρξει μια νέα συμφωνία η οποία να βελτιώνει την υπάρχουσα κατάσταση και ε, τη συμφωνία, την πρόταση αυτή θα την στείλουμε εδώ, θα την υπογράψουμε στις Βρυξέλλες σε λίγους μήνες. Θα ήθελα να πω επίσης ότι το Eurojust εμπλέκεται επίσης σε 12 αναλυτικούς φακέλους έρευνας τα δύο τρίτα δηλαδή ε, των προτάσεων που είχαν γίνει έχουν ήδη ανοίξει και είναι υποδιερεύνηση. Συνεργαζόμαστε και με χώρες μη μέλη όπως την Κροατία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νορβηγία κτλ. Υπογράψαμε το 2008 μια συμφωνία συνεργασίας με την Ελβετική Συνομοσπονδία, είναι βασικός μας εταίρος, όπως επίσης και με τη Φιρόμ. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας και με, μια διεθνή οργάνωση η οποία έχει σημεία επαφής δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας της Λατινικής Αμερικής, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας. Η συνεργασία με την Ισπανία είναι πάρα πολύ σημαντική σε συγκεκριμένους τομείς όπως τα ναρκωτικά. πέντε σημεία θα ήθελα να σημειώσω που είναι σημαντικά για το Eurojust και τις μελλοντικές εξελίξεις του Eurojust. Αυτό είναι θα έλεγα βασικό στόχος και των κρατών μελών και του Eurojust και για τα εθνικά κοινοβούλια. Πρέπει αυτές τις αποφάσεις να τις εφαρμόσουν. Πέντε σημεία λοιπόν. Το πρώτο έχει σχέση με την με το θέμα της εσωτερικής λειτουργίας του Eurojust, με το καθεστώς των κρατών μελών στο εσωτερικό του Eurojust. Θα πρέπει να μπορούν στο εσωτερικό της Eurojust οι χώρες να λειτουργούν σωστά. Γιατί πάρα πολύ συχνά κάποια μέλη από χώρες δεν είναι μόνιμοι θα έλεγα συνεργαζόμενοι με το Eurojust. Υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες δεν είναι παρούσες μονίμω στη Χάγη. Απλώ έρχονται, ενεργούν από του χώρε και έρχονται στη Χάγη μόνο για κάποιες συνεδριάσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα μπορέσει να διευθύνει αυτό το πράγμα εκ μέρου των κρατών μελών. Τι μπορώ να σας πω, το 50% των κρατών μελών δεν έχουν ε, ε, αντιπροσώπους, αναπληρωτές ή ε, βοηθούς 6 χρόνια μετά την δημιουργία, 7 χρόνια μετά τη δημιουργία της Eurojust. Επίσης, Πρέπει να πω ότι βασικά οι αρμοδιότητές μας είναι οι ίδιες, αλλά όλο και περισσότερο αναγνωρίζεται ο ρόλος μας, διότι βοηθούμε όλα τα εθνικά καρμαθητικά συστήματα. Πρέπει όμως όλοι να αναγνωρίσουν την Eurojust. Διαφορετικά δεν μπορούμε να ενεργήσουμε σωστά. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών. Εμείς δεν παράγουμε πληροφορία, δεχόμεθα πληροφορίες και χειριζόμαστε τις πληροφορίες οι οποίες φτάνουν στα χέρια μας από τα κράτη-μέλη και πρέπει να προσφέρουμε και προσφέρουμε τις συνθήκες που χρειάζεται για να προστατεύονται αυτές οι πληροφορίες σε θέματα ποινικά. Έχουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια φτιάξει ένα ε, σύστημα τέτοιο που να μας επιτρέπει να προστατεύουμε τέτοιου είδους δεδομένα. Επίση είναι σημαντικό ο ρόλο μα στην εργασία με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, με τι εθνικέ αρχέ. Έχουμε το τομέα τη δικαιοσύνη. Αλλά πολλές χώρες δεν διαθέτουν ούτε καν γραμματεία για να υποβοηθηθεί στο έργο που κάνουμε εμείς. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια νέα απόφαση βάσει της οποίας θα μπορέσουν να λειτουργήσουν τα διάφορα δίκτυα όπως το δίκτυο για τις κοινέ ερευνητικέ ομάδες, ε, για την ε, ε, διαφθορά, για τις γενοκτονίες. Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω είναι η σύσταση εθνικών συστημάτων συντονισμού. Δεν μπορούμε να κάνουμε συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν δεν υπάρχει συντονισμός όλων των αρμοδίων οργάνων σε εθνικό επίπεδο. Η επόμενη παρατήρηση αφορά τη σχέση μας με τη Frontex. Έχουμε υπογράψει με την Interpol, με το CITSEN και με τη Frontex διάφορες συμφωνίες. Τελειώνοντας θα σας αναφέρω τα θέματα τα οικονομικά, τον προϋπολογισμό. Οι ανάγκες μας όλο και μεγαλώνουν. Το 2008 πήραμε 20 εκατομμύρια και στον διορθωτικό προϋπολογισμό πήραμε άλλα 4,8. Το 2009 θα ξεστεί αυτό το ποσό. Ζητήσαμε ε, συμπληρωματικό ποσό στον προϋπολογισμό. 3 εκατομμύρια ευρώ. Εκρεμεί ακόμη η έγκριση αυτού του συμπληρωματικού ποσού και ελπίζουμε ότι θα ακούσουμε τα καλά νέα σύντομα. Και για το 2010 ε, έχουμε ζητήσει 33 και φαντάζομαι ότι θα υπάρξει περικοπή στα 30 εκατομμύρια. Συμπεραίνοντας, θα ήθελα να πω το εξή. Πιστεύουμε ότι εμείς στη Eurojust ότι η δημιουργία της Eurojust είναι ορόσημο στην προσπάθεια να δημιουργήσουμε έναν ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Έχουμε εργαστεί μέχρι τώρα στο μίσ που μας αφορούν πάρα πολύ σκληρά, κάνουμε τις αιτήσεις αναφορές μας. Ελπίζουμε ότι η δουλειά που κάνουμε είναι, ε, έχει προστιθέμενη αξία στην καταπολέμηση του διαμεθοριακού εγκλήματος και βεβαίω ξέρουμε ότι πάντα έχουμε την υποστήριξή σα. Εμπιστοσύνη ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε την υποστήριξή σα. Καλή συνεργασία. Κάτι άλλο το οποίο πρέπει να πω είναι ότι θα πρέπει να είμαστε και επικριτικοί για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε επίσης σε θέματα ε, διαδικασιών που ακολουθούμε για την καταπολέμηση του διαμεθοριακού κλίματος. Θα ήθελα τελικά να ευχαριστήσω την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την ε, γνωμοδότησή της που αφορά τη νέα απόφαση που αφορά τη Eurojust. Ήδη κάποιους εκπροσώπους τους συναντήσαμε στη Χάγη. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να την χάνουμε τη υποστήριξή σας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα είμαι έτοιμος να ακούσω τις ερωτήσεις σας. Εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε για την παρουσίαση της 7 η ετησίας έκθεσης. Έχουμε πέντε συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Σας εκλυπαρώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Να σεβαστείτε το χρόνο που σας δίνω. Ένα λεπτό ο καθένας. Όχι παραπάνω. Για να μπορέσουμε να τελειώσουμε έγκαιρα και να σεβαστούμε και τον χρόνο εργασία των διερμηνέων. Η κυρία Μπόσκουτ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι οι δραστηριότητες της Eurojust αυξάνονται βλέπουμε πόσες εκατοντάδες υποθέσεων απάτης ή παραπτωμάτων εξετάστηκαν από τη Eurojust. Έχουμε εδώ να κάνουμε με θέματα τα οποία αφορούν διάφορες χώρες δικές μας. Δεν βλέπω όμως να αναφέρονται απάτες που αφορούν κονδύλια που χρησιμοποιούν Ισλαμικές οργανώσεις. Και ξέρουμε ότι φορές Κάποιες φορές ε, χρησιμοποιούνται τα, οι περίφημες πυραμίδες, οι οποίες ε, ε, έχουν οδηγήσει στην οικονομική καταστροφή πολλά χιλιάδες άτομα. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στη χώρα μου. Και όχι μόνο, αλλά και σε άλλες χώρες. Και υπάρχει μια υποψήφια χώρα που δεν κάνει τίποτα για αυτό το θέμα αυτό. Γιατί δεν σας ενδιαφέρουν τέτοιου υποθέσεις. Ο κύριος Λέλο. Ευχαριστώ κύριε Λόπες Δαμότα για αυτά που είπατε. Ξέρω ότι εσείς συντονίζετε τις δραστηριότητες των ε, καστικών αρχών. Σε αυτή τη στιγμή στην ε, Πορτογαλία ζητήθηκε από την Eurojust να γίνει έρευνα σε μια πάρα πολύ σημαντική εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετέχουν ε, δημόσια πρόσωπα και όπου μπορείτε εσείς να διαδραματίσετε αναπτύσσεται πολύ σημαντικό ρόλο και ως Πορτογάλος. Όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή γίνεται κάποια έρευνα για την ε, προσπάθεια ενδεχομένως να ασκήσει κάποιος επιρροή στην εκδίκαση και στην εξέταση μιας ε, απόφαση στην οποία έχουν δικαστικές αρχές Αγγλίας και Πορτογαλίας. Εγώ στα πλαίσια της ετήσιας έκθεσης του 2008 γιατί δεν μας αναφέρετε τέτοιου είδους υποθέσεις όπως αυτής. Φαντάζεστε ότι δεν δικαιολογείται. Μήπως θα πρέπει να υποφεληθεί η Πορτογαλία από τη δική σας παρουσία ε, στη Eurojust για να βοηθηθεί και να ενεργήσει πιο αποτελεσματικά. Ο κύριος Δία Δεμέρα, ένα λεφτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Eurojust για την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσής σας. Ένα σχόλιο και μια ερώτηση. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσετε τα ευάλωτα σημεία της Eurojust. Πρόκειται για ένα παιδάκι 6 ε, ετών που έχει αυξημένες ε, ανάγκες διατροφής, αλλά βλέπω ότι τρέφεται σωστά και μεγαλώνει σωστά. Πρέπει να σας πω ότι κάνετε κάποια πράγματα τα οποία ε, κάνει και η Όλαφ και η Europol. Στην ετήσια έκθεση λέτε ότι το 2008 είχατε για τη δική μας, για τις διάφορες ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28 ε, αιτήσει ε, Ε, σύλληψης η οποία δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί δεδομένου ότι δεν υπήρχαν τα κατάλληλα στοιχεία. Μήπως μπορείτε εσείς να βελτιώσετε τα πράγματα. Κυρία Λούτφορντ, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση κύριε Πρόεδρα. Στην ετήσια έκθεση το πλεονέκτημα είναι ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία. Το μειονέκτημα ότι δεν διαβάζουν όλοι. Θα ήθελα να υπάρχει περισσότερη λεπτομέρεια στα θέματα που αναφέρει σελίδες 30 και 31. Ε, προσκόμματα σε θέματα συνεργασίας. Επίσης, είπατε ότι σε θέματα ε, χρηματοδότησης τραμοκρατών και στα κονδύλια τα, τα οποία υποφελούνται υπάρχει καθυστέρηση δύο ετών. Θα πω λοιπόν αντίθετα με τον κύριο Δίας Δεμέρα ότι η πολιτική βούληση και οι αποτελεσματικές κυβερνητικές αποφάσεις μπορεί να οδηγήσουν στην ε, ε, αποτελεσματική εφαρμογή κάποιων μέτρων, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις καθυστέρησης και παραβιάσεων. Ξέρω ότι έχετε προβλήματα και προορισμού, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει περισσότερο τα στοιχεία με τα οποία ασχολείστε, τα θέματα που αφορούν ε, το SWIFT, τις βασικές, ε, ε, το PNR, τέτοιου είδου θέματα, να την χάνουν καλύτερε έρευνε. Και δεν μπορείτε να κάνετε περαιτέρω έρευνε σε τέτοιου είδου θέματα, δεδομένου ότι δεν έχετε πάρα πολύ, πολλά κονδύλια. Βεβαίω, το θέμα της ασφάλειας των συνόρων είναι σημαντικό, αλλά το θέμα της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται να είναι δευτερεύουσα σημασία. Και αν δεν γίνεται η σωστή έρευνα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και βεβαίως θα πρέπει να αναφέρονται όλες τις περιπτώσεις στις οποίες έχουμε ε, ε, για βασικά τέτοιου είδους θέματα ή καθυστέρηση στην έρευνα ή μη ε, ανταλλαγή κάποιων βασικών δεδομένων. Κύριε Βέμπερ, σας ευχαριστώ κύριε Μότα για τη δουλειά που κάνετε στην Eurojust, την υποστηρίζει, διότι πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια αποδείξατε ότι πρόκειται για έναν οργανισμό τον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε και στον οποίο μπορούμε να δώσουμε περισσότερες αρμοδιότητες από ό,τι σήμερα. Πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη έχουν κάποιους ενδιασμούς. Δεν θέλουν να σας δώσουν ε, πολλές εξουσίες για να κάνετε τη δουλειά σας. Ως μαρτυρία είναι ότι η απόφαση της 4ης Ιουνίου μετά από την τρομερή άσκηση, ε, πίεση που μας ασκήθηκε ακόμη δεν έχει στεθεί σε εφαρμογή. υπάρχει το θέμα της ε, ε, διαμάχες που μπορεί να υπάρξει εξαιτίας των ε, διαφορετικών δικαιοδοτικών οργάνων και προβλημάτων που μπορούν να, προβλήπ, να προκύψουν. Υπάρχουν κάποιες χώρες μία έως πέντε που ίσως δεν ενεργούν σωστά. Ίσως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται να έχουν ε, περισσότερη σχέση με σας. Είναι διότι έμαθαν πιο πολλά μέχρι τώρα και έχετε καλύτερη συνεργασία μεταξύ του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χουάρεγγε για ένα λεπτό. Η ειλικρίνεια των ε, παρεμβάσεων σας νομίζω ότι μας επιτρέπει να κάνουμε μια κριτική για σας. Πρόκειται για μια τρομερή ιδέα που υπήρχαν αυτοί που έκανε τη Eurojust, αλλά δεν δουλεύει το σύστημα. Οι στατιστικές είναι πολύ φτωχές. Υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές χώρες όπως η Γαλλία ή το Ηνωμένο Βασίλειο που μείωσαν τις στατιστικές τους από ό,τι βλέπουμε. Είχαν περισσότερες περιπτώσεις που έφτασαν σε το 2007 παρά το 2008. Μας είπατε επίσης ότι κάποια μέλη δεν έχουν εκπροσώπους στη Χάγη, δεν παίρνουν τις πληροφορίες, δεν θέλουν να συνεργαστούν και πραγματικά πρέπει να σας πω ότι έχω μεγάλη απογοήτευση αισθάνομαι για το πώς δουλεύει η Eurojust. Η ιδέα είναι πραγματικά ευφυής, και νομίζω ότι θα πρέπει η Κομισιό να αναθεωρήσει και το οργανόγραμμά σας ή μάλλον η δική μας Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ζητήσει από την Εκτελεστική Επιτροπή να κάνει αναθεώρηση του τρόπου τον οποίο σκέπτεται το όργανο του οποίου ηγείστε. Το οργανόγραμμά σας επαναλαμβάνω, τις αρμοδιότητές σας, το ρόλο σας, να κάνει αξιολόγηση δουλειά που έχετε κάνει και των κονδυλίων που σας δίνει για να γίνετε καλύτεροι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε το συντομότερο δυνατό. Παρακαλώ να απαντήσετε σε 7 λεπτά το αργότερο. Ευχαριστώ. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με τα κονδύλια των ε, Ισλαμικών οργανώσεων, όπως είπε η κυρία Μποσκούρ. Το ερώτημα είναι γιατί αυτό το θέμα δεν είναι από τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε. Είναι πολύ απλή η ερώτηση, η απάντηση στην ερώτηση αυτή. Ενεργούμε εάν μας το ζητήσει κάποιο κράτος μέλος. Εάν κάποιο κράτος μέλος δεν μας ζητήσει να παρέμβουμε και να κάνουμε κάτι, δεν κάνουμε τίποτε. Και δεν ξέρουμε τίποτα για τέτοιου είδους περιπτώσεις. Αυτό λοιπόν που μπορώ να σας πω είναι ότι όταν μας ζητείτε να κάνουμε κάτι από κάποιο κράτος μέλος, κάνουμε, ενεργούμε. Εάν κάποιος δεν μας ζητήσει να κάνουμε κάτι, δεν κάνουμε τίποτε. Δεδομένου ότι δεν έχουμε νομική βάση που θα μας το επιτρέπει. Περιμένουμε λοιπόν να υποβάλει έτοιμα μία ερώτηση και στη συγκεκριμένη αυτή περίπτωση δεν ξέρω γιατί εγώ δεν έχω, αν θέλετε, ως εθνικό μέλος Πορτογαλίας εξαιτία των θεμάτων προστασία των προσωπικών δεδομένων πρόσβαση σε θέματα που δεν αφορούν τη χώρα μου, αλλά μπορώ να σας πω ότι εάν το θέμα αυτό είναι ένα θέμα με το οποίο δεν ασχολείται η Eurojust, γιατί κανένας δεν μας έκανε αναφορά περί τούτου κάποιοι που πιστεύουν ότι δεν χρειάζονται τη Eurojust. Γιατί για να πάει κανείς στη Eurojust σημαίνει περισσότερη δουλειά και για τι αγγελικές αρχέ και για τι ε, αστυνομικέ αρχέ που ασχολούνται με ένα θέμα σε εσωτερικό επίπεδο και ίσω δεν έχουν περισσότερου πόρου να στείλουν στη ΧΑΗ για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Επίση, κάποιοι πιστεύουν ότι καλύτερα να ασχοληθούν με την παραχάραξη ή με την πλαστογράφηση ενός εγγράφου με το ίδιο το έγγραφο, ένα διαβατήριο Φερρυπίν, παρά να το να ψάξουν να βρούνε αυτοί που το πλαστογράφησαν ποιοι είναι και πού είναι. Κύριε Ντεμέλο, θα σας μιλήσω στο τέλος πορτογαλικά για να σας απαντήσω το ερώτημά σας. Τώρα, σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Κύριε Ντίας Δεμέρα, Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα στο τομέα αυτό. Υπάρχει ένα μοντέλο, αν θέλετε, που έχει δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα, αλλά πολλές φορές οι εθνικές αρχές αποφασίζουν να είναι δημιουργικές και να παρουσιάσουν, αν θέλετε, το layout με διαφορετικό τρόπο. Και έτσι όταν δεν είναι κάτι ομοιόμορφο δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Καθυστερούμε. Πολλές φορές δεν γίνεται ακόμη σεβαστή και η αρχή της ε, ειδική περίπτωση αυτής. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας ε, ανάκρισης βλέπουμε ότι στη το ένταλμα έχει εκδοθεί για ένα συγκεκριμένο αδίκημα παράπτωμα έγκλημα και υπάρχουν κι άλλα. Πολλές φορές λοιπόν έχουμε τέτοιες δυσκολίες, μπλέκονται τα πράγματα και πολλές φορές καθυστερούμε και είναι και πολύ αργά. Αλλά θα μπορούσα να σας πω ότι συνήθως επιλύουμε τέτοιου είδους προβλήματα και ξεπερνάμε τέτοιου είδου δυσκολίε. Αλλά δεν συνηθίζει κανείς να συμβουλευτεί ούτε τη Eurojust ή τις άλλες ε, δικαστικές αρχές πριν να εκδοθεί το ευρωπαϊκό ε, ένταλμα σύλληψης. Και πολλές φορές έχετε δύο ε, αρχές οι οποίες εκδίδουν το ίδιο ένταλμα σύλληψης για το ίδιο άτομο. Και καμιά φορά επιλαμβάνονται τις υπόθεσεις δύο διαφορετικοί δικαστές, ο ένας λέει ναι, ο άλλος λέει όχι και καταλήγουμε σε ένα χάος. Και πολλέ φορέ όταν φτάνουν τέτοιου είδου θέματα στη Eurojust, καταλήγουμε συμφωνίε και βρίσκουμε λύσει. Αλλά όντω, πολλά πρέπει να γίνουν για να μην εκκρεμούν τέτοιου υποθέσει, να μην καθυστερούν και σε σχέση με την, εφαρμογή. Κυρία Λάντφορντ, όντως είναι απογοητευτικό πολλές φορές να βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν εφαρμόζεται σωστά στις διάφορες χώρες. Κάποιος έγραψε σε ένα βιβλίο ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τρίτο πυλώνα είναι εικονική. Ελπίζω ότι με την ε, θέση σε ισχύ της Συνδίκης Λισαβόνας θα αλλάξουν τα πράγματα διότι πρέπει να σας πω ότι η απόφαση για τη Eurojust εγκρίθηκε το 2002 και υπήρχε υποχρέωση των κρατών μελών μέχρι το Σεπτέμβριο 2003 να μεταφέρουν ε, την απόφαση στο εθνικό τους δίκαιο. Ξέρετε πόσες το έκαναν, μία χώρα, μία και μοναδική. Η Πορτογαλία, αν μου επιτρέπετε να το πω. αλλά μόνο 50% των κρατών μελών έχουν μεταφέρει, μάλλον έχουν εγκρίνει από την νομοθεσία. Πράγμα που σημαίνει ότι 13 ή 14 ακόμη δεν έχουν εγκρίνει τη σχετική νομοθεσία ε, για την μεταφορά της απόφασης που αφορά το, την δημιουργία της Eurojust από το 2002. Η Ισπανία, Φερρυπίν κύριε Χουάρεγγι. Το έκανε αυτό το 2006. Το 2006. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ισπανία είναι μία από τις χώρες που παρουσιάζει τις περισσότερες ε, υποθέσεις στη Eurostat, εκατοντάδες υποθέσεων. Και κοιτάξτε εδώ, πόσες χώρες είναι αυτές οι οποίες προστρέχουν στην Eurojust. Η Ισπανία δεν ε, στέλνει θέματα στη Eurojust. Η Eurojust αντιθέτως προσφεύγει πολύ συχνά στην Ισπανία. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ε, υποθέσεις που φτάνουν σε μας. Αλλά πρέπει να σας πω ότι τώρα ε, έχουμε και εκπροσώπηση στη Eurojust της Ισπανίας. Για 5-6 χρόνια είχαμε μόνο έναν εθνικό εκπρόσωπο αποσπασμένο και κάνουμε τη δουλειά μας με ένα άτομο. Και χρειάστηκε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα αυτό κάνοντας πρόσφυγη και στον Υπουργό και στον ε, Γενικό Εισαγγελέα διότι είχαμε έναν ε, κακομύρι ο οποίος κάθε εβδομάδα σαν ποδοσφαιριστής πήγαινε και ερχότανε για να μπορέσει να χειριστεί τις υποθέσεις που αφορούσαν τη χώρα. Εν πάση περιπτώσει τώρα άλλαξαν τα πράγματα και έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Και θα ήθελα να συγχαρώ την Ισπανία γι' αυτό που έκανα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα είμαστε φτωχοί αν θέλετε. Έχουμε λίγες, ε, λίγα κονδύλια στη θέση μας, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Διαβάζοντας την εκθεσή μας θα δείτε πολλά ενδιαφέροντα μέσα. Και πρέπει να πω ότι είμαστε η μοναδική οργάνωση στον κόσμο που ασχολείται με τέτοιου είδους ε, υποθέσεις και έχουμε κινήσει το ενδιαφέρον και πολλών αρχών εκτός Ευρώπης. Και βεβαίως κάνουμε ό,τι μπορούμε με τις περιορισμένη οικονομική ενίσχυση που παίρνουμε από τις διάφορες χώρες μέλη. Ευχαριστώ την κυρία Βέμπερ για τα ευγενικά της λόγια. Είχαμε την δυνατότητα να συζητήσουμε κάποια θέματα και είσαστε είχατε τη δυνατότητα να έρθετε στη Euro Just να σας κάνουμε μια παρουσίαση και εσάς και συναδέλφους σας είπαμε δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Έτσι είναι η Eurojust. Ρωτήστε μας ό,τι θέλετε να σας πούν τα πάντα. Κοιτάξτε παντού ό,τι βλέπετε είναι η κατάσταση που υπάρχει. Ξέρω ότι είσαστε υπεύθυνοι για την γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να πω ότι μας χαροποιεί ιδιαίτερω η γνωμοδότηση. Ο κύριος Νούνο Μέλο τώρα. Πρέπει να σας πω ότι περίμενα να μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Όταν μπήκα στην αίθουσα και σας είδα, είπα, ο κύριος Νούνοντε Μέλο θα είναι εδώ για να μου κάνει μόνο αυτή και την μοναδική ερώτηση. Δεν με ρωτήσατε τίποτα για την Eurojust. Κύριε Βουλευτά, εγώ πρέπει να σας πω το εξής. Εσείς αναφερθήκατε σε ένα θέμα εθνικό δικό μας, πορτογαλικό. Εγώ δεν έχω ως πρόεδρος της Eurojust να πω τίποτε. Τα θέματα τα εθνικά συζητούνται στην Πορτογαλία και όχι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως πρόεδρος της Eurojust, κύριε Βουλευτά, θα πρέπει να πω το εξής. Ότι έχω την πλήρη υποστήριξη της Eurojust με εξέλεξαν οι συνάδελφοί μου, δεν με διόρισε το πορτογαλικό κράτος. Η Πορτογαλία δεν έχει να κάνει τίποτε με την δική μου θέση ως Προέδρου της Eurojust. Δεν θέλω ε, να μην είμαι ευγενής. Θα ήθελα να απαντήσω το ερώτημά σας. Γιατί είπατε ότι εγώ δεν ενημέρωσα και γιατί ανέστηλα την όλη υπόθεση αυτή. Θα πω το εξή. Η Πορτογαλία δεν πάει στο Eurojust. Την αποφεύγει. Διότι υπάρχει κάποιο προσωπικό θέμα. Εάν δείτε εδώ, η Πορτογαλία είναι μεταξύ των πέντε καλύτερων χωρών που προσφεύγουν στη Eurojust. Τώρα, στην υπόθεση αυτή Freeport, για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση την οποία ε, αναφέρεστε. Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξή. Η Πορτογαλία δεν ζήτησε ποτέ την υποστήριξη της Eurojust. Η διαδικασία άρχισε το 2004-2005 στην Πορτογαλία. Η Πορτογαλία ποτέ δεν ζήτησε την υποστήριξη της ε, Eurojust για οποιαδήποτε συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εισαγγελική παραγγελία Συγγνώμη, συγγνώμη, να μην με ακρηγορείτε, λέει ο πρόεδρο. Λοιπόν, η επιστολή αυτή έστειλε, στάλει το 2005 το Ηνωμένο Βασίλειο, ποτέ δεν μας ενημέρωσε κανείς και τρία χρόνια μετά ήρθε το Ηνωμένο Βασίλειο να μας ζητήσει τη δική μας συνδρομή, διότι η Πορτογαλία δεν είχε δώσει σε αυτή την επιστολή καμία απάντηση. Εμείς λοιπόν μπήκαμε σε όλη αυτή τη διαδικασία ετήσι του Ηνωμένου Βασιλείου. Με αυτή, ασχοληθήκαμε με αυτή την υπόθεση για έξι μήνες. Και το Μάρτιο του 2000 αφού κάναμε δύο συντονιστικές συναντήσεις, ε, τις οποίες πληρώσαμε, καταβάλαμε δηλαδή όλα τα έξοδα, και μετά από ανταλλαγή πληροφοριών και αφού ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα, τελικά ο Άγγλος συνάδελφος πρέπει να σας πω ότι αποφάσισε να κλείσει την υπόθεση το Μάρτιο του 2009. Κατά συνέπεια, η Πορτογαλία ποτέ δεν ζήτησε τίποτα στη Eurojust, ούτε πριν ούτε μετά. Άρα, επαναλαμβάνω, δεν ε, πήγε η Πορτογαλία, δεν ήρθε μάλλον η Πορτογαλία σε εμά στη Eurojust. Δεν θα ήθελα να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. Επαναλαμβάνω, ποτέ για αυτό το θέμα δεν ήρθε η Πορτογαλία στην, ε, στο Eurojust. Έγινε η έρευνα από τη μεριά της ε, Ηνωμένου Βασιλείου που αποφάσισε μετά από εξέταση του όλου θέματος για έξι μήνες να κλείσει την υπόθεση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κλείσει το θέμα αυτό. Βλέπω όμως ότι υπάρχουν άλλοι δύο συνάδελφοι που έχουν ζητήσει το λόγο. Μόνο εφόσον θεωρείτε ότι άπτεται άμεσα με το συζητούμενο θέμα, τότε να περιοριστείτε σε 50 δευτερόλεπτα. το θέμα αφορούσε, θα έλεγα, μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Γι' αυτό θα συνεχίσω πορτογαλικά. Κύριε Μπότα, εγώ δεν ήθελα να συζητηθεί το θέμα αυτό της ανακριστικής διαδικασίας. Ήθελα να συζητηθεί το θέμα της συνεργασίας μεταξύ όλων των κρατών, όπως και η Πορτογαλία, με τη Eurojust. Είπατε εσείς ε, ότι έπρεπε να συζητηθεί αυτό στο Πορτογαλικό Κοινοβούλιο. Εγώ προσπάθησα να το κάνω, αλλά δεν με άφησαν οι σοσιαλιστές στην Πορτογαλία. Γι' αυτό το ανέφερα εδώ. Κύριε Λόπες Δεμότα, μπορείτε να μιλήσετε με τον συντενιστή, τον κύριο Κέρκοφ για θέματα τρομοκρατίας, γιατί στην έκθεση του Ιουνίου λέει ότι όλα τα κράτη-μέλη, εκτός από τη Βουλγαρία, έχουν... Ε, ε, ε μεταφέρει και έχουν εγκρίνει την ε, απόφαση πλαίσιο. Θα ήθελα λοιπόν ε, να τσεκάρετε τα δύο έγγραφα για να δούμε ποιο από τα δύο λέει την αλήθεια. Ο κύριος Ντοκέρκοφ θα έρθει αύριο. Έγγραφο της Δευτέρας Ιουνίου είναι αυτό το, στο οποίο αναφέρομαι. Έγγραφο του Συμβουλίου για την εφαρμογή του σχεδίου για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας. Είναι το έγγραφο για το οποίο θα μας μιλήσει ο κύριος Δεκερκόβ. Όχι, όχι, όχι, όχι. Την απόφαση για, την, ε, για τη Eurojust, για την τρομοκρατία. Πράγμα σημαίνει ότι πολλοί δούλεψαν σωστά το 2009. Όταν ενέκρινε την απόφαση στο Συμβούλιο το 2008, Αυτά τα στοιχεία είχα εγώ. Το 50% των κρατών μελών δεν την είχαν εφαρμόσει. Αλλά ευχαρίστως να σας δώσω όλα τα στοιχεία τα σημερινά. Αλλά χαίρομαι που υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Ακούστε, εγώ μιλάω για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητο έχει τεθεί αυτό και στην πράξη. Ακούστε. Εγώ δεν θα αφήσω τη θέση μου, ούτε θα παραιτηθώ. Δεν έχω κανένα τέτοια πρόθεση, διότι δεν υπάρχει βάσιμος λόγος από νομική πλευρά. Δεύτερον, η Eurojust με εμπιστεύεται πλήρως και με πολύ μεγάλη τιμή, ευχαρίστηση και υπερηφάνεια εκπροσωπώ ως πρόεδρος Eurojust τον οργανισμό μου. Ασχολούμαι με το θέμα αυτό εδώ και δέκα χρόνια. Πρέπει να σας πω ότι και εγώ ασχολήθηκα με την ε, πολιτική. Ασχολούμαι τη Eurojust εδώ και χρόνια. Τη θεωρώ λίγο το παιδάκι μου. Και αισθάνομαι υπεύθυνο για την Eurojust. Και ω πρόεδρο τη ομάδα μου και ω αντιπρόεδρο τη Eurojust και ω πρόεδρο έχει αναγνωριστεί η εργασία την οποία επιτελώ. Αναγνωρίζω τη σημασία που έχει συνεργασία με του συναδέλφου. Αναγνωρίζω την υποστήριξή του. Και πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ περήφανη αυτό που κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ε, παρουσία σας, την παρουσίασή σας και εύχομαι τα καλύτερα για την περαιτέρω εξέλιξη της οργάνωσης που ήρθατε σήμερα να μας παρουσιάσετε. Ευχαριστώ. Ε, ε, I think we should... Νομίζω ότι τώρα θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο αυτό το οποίο αναβάλαμε σήμερα το πρωί να συζητήσουμε αφορά τη διαδικασία προϋπολογισμού για το 2010 με τιμά ο διορισμός μου σαν εισηγητή θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τα βασικά στοιχεία της πρότασης την οποία σας υπέβαλα την προηγούμενη εβδομάδα και μετά θα ξεκινήσει η συζήτηση για να μπορέσω να πάρω και τις δικές σας πρώτο τροπολογίες και σε σχέση με τις γραμμές του προϋπολογισμού και σε σχέση με τη γνωμοδότηση. Θα μιλήσω ισπανικά. Είναι σαφές ότι οι τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί στην αρμόδια επιτροπή και που περιλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης αναφορικά με το προσχέδιο του προϋπολογισμού. Ε, εξετάστηκαν σε βάθος οι τροπολογίες αυτές έτσι ώστε να αποκατασταθεί θα έλεγα η ισορροπία που χαρακτήριζε τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Τώρα θα αναφερθώ ειδικά στα θέματα που αφορούν τις ελευθερίες, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια και ότι έχει σχέση και με τις ανεξάρτητες αρχές, ευρωπαϊκές αρχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κτλ. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού είχαν ληφθεί ορισμένες αποφάσεις οι οποίες οδηγούν σε μία αύξηση κατά 3,5% σε σχέση με τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Σχετικά τώρα με την πολιτική θεωρήσεων τα εξωτερικά σύνορα, θεμελιώδη δικαιώματα, το 18-4 δηλαδή, τα θέματα δικαιοσύνης έχει υπάρξει μια αύξηση 4,7% και 3, 37% σε σχέση με το 2009. Στο κεφάλαιο ε, ελευθερίες αυξάνεται κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό ο προϋπολογισμός ε, σε σχέση με το 2009 λόγω της ένταξης νέων μέτρων στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Εν πάση περιπτώσει, το κεφάλαιο το σχετικό με τη μετανάστευση μειώνεται κατά 1,50%. Κάτι το οποίο δεν μας αφήνει ικανοποιημένους. Τα στοιχεία υποστήριξης στους ε, πρόσφυγες και το σχέδιο για την ένταξη της Ευρωπόλ στα κοινοτικά όργανα βλέπουμε ότι υπάρχουν ορισμένα προβλήματα. προσωπικά θα έλεγα ότι η δημοσιονομική πρίκα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ανεπαρκής. Εμείς είμαστε φυσικά διατεθειμένοι να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περαιτέρω ενίσχυση δημοσιονομική. Ακόμα και σε περιπτώσεις όπως το Frontex. Ο Αλβάρο και Γκρίσμπεκ προτείνουν μια αύξηση των πιστώσεων πληρωμών. Είναι κάτι το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει να υπάρξουν βασικές μεταφορές κατά τη διάρκεια του 2010 αν χρειαστεί αυτό. Ο κύριος Μπουσούτιλ. και αυτός μια αύξηση του προϋπολογισμού για το Frontex την οποία σας την υποβάλλω στα πλαίσια της ε, πρότασής μου σχετικά τώρα με το Ταμείο για τα Εξωτερικά Σύνορα. Έχουμε τροπολογία της κυρίας Χένης Πλέσσερ. Συμφωνούμε με την τροπολογία αυτή. Εμείς ναι, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ακούσουμε και τι έχει να μας πει η Κομισιόν. Επίσης υπάρχουν οι τροπολογίες του κυρίου Τζακολίνο που αφορούν τις ενισχύσεις τα κράτη των κρατών μελών για τους πρόσφυγες και τους ετούντες άσυλο. Ο παρόν μηχανισμός φαίνεται ότι μάλλον ευνοεί τις χώρες που είναι η πρώτη αποδοχής των προσφύγων και των ετούντων άσυλο και πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει επίσηγουσα ανάγκη τη αιτήση των κρατών μπορούν να χορηγηθούν για να βοηθηθούν οι πρόσφυγες και κάποια επίγουσας φύση κονδύλια. Κύριο Τζακολίνο λέει ότι μετά από την κατάλληλη Ε, νομική ε, γνώμη την οποία ζήτησε ότι αυτό το θέμα είναι ένα θέμα το οποίο αφορά και τροπολογία που κατέθεσε ο κύριος Μπουσούτιλ και ο κύριος το θέμα αυτό φαίνεται ότι συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό. Λαμβάνοντα υπόψη πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό, θα πρέπει να ακούσουμε και την ε, Κομισιό, αλλά πιστεύω ότι η έκθεση της Επιτροπής θα πρέπει, η αναφορά μάλλον, η γνωμοδότηση της Επιτροπής για αυτό το θέμα να συμπεριληφθεί στις ε, τροπολογίες. Εμείς είμαστε υπέρ αυτής της τροπολογίας. Τώρα, σε περίπτωση μαζικής ε, άφηξης προσφύγων υπάρχει ένα ειδικό θέμα που αφορά την ε, Child Protection Reallocation, την ε, χορήγηση κάποιων κονδυλίων για τα προστασία των παιδιών. Είμαστε υπέρ της συμβαστικής τροπολογίας αυτής. Επίσης αναφέρεται κάτι σε σχέση με βοήθεια προς τρίτες χώρες, τροπολογία του κυρίου Κροσέτ, όλα αυτά που αναφέρονται για να ενισχυθεί ο διάλογος, η επικοινωνία, οι γλώσσες, τα προγράμματα, τα εκπαιδευτικά και τα πολιτιστικά για να μπορέσουν να ενσωματωθούν καλύτερες κοινωνίες προερχόμενα άτομα από τρίτες χώρες, ε, μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε ποια είναι η άποψη της Κομισιόν. Κάποια άλλη τροπολογία αφορά την πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητα. Την πρόληψη σε θέματα ε, λαθρεμπορίων ναρκωτικών. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακούσουμε την Κομισιόν δεδομένου ότι τέτοιου είδους θέματα συμπεριλαμβάνονται και σε άλλες γραμμές του προπολογισμού. Υποστηρίζουμε την τροπολογία που αφορά την διαφάνεια που προτείνεται μεταξύ άλλων από τον κύριο Κάσμαν και την τροπολογία που αφορά τους εξαφανιστέντες στην Κύπρο, τους αγνοούμενους στην Κύπρο. Με αυτή τη συνοπτική παρουσίαση που έκανα αρχίζει η συζήτηση για να δούμε ποια είναι η γνώμη των διαφόρων ομάδων πριν να κάνουμε την ε, οριστική παρουσίαση της έκθεσης αυτής. και να παρουσιάσουμε τις ε, τροπολογίες με προθεσμία την 7η Σεπτεμβρίου. Ποιος θέλει το λόγο παρακαλώ. Ο κύριος Μπουσούτιλ. Θέλετε κύριε Μπουσούτιλ να πείτε κάτι. Ναι, πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε για την παρουσίαση και της γνωμοδοτησής σας αλλά και την αξιολόγηση των τροπολογιών. Πολύ σύντομα λοιπόν, εξ ονόματος του Λαϊκού Κόμματος. Και σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότησή σας, συμφωνούμε, υποστηρίζουμε τα θέματα που θίγεται. Εδώ θα αναφέρω δύο σχόλια. Πρώτο, σε ό,τι αφορά την Frontex. Και αν κατανοώ σωστά, στη γνωμοδότησή σας λέτε ότι ε, θα πρέπει να παραμείνει ο προπολογισμό τη στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Υπενθυμίζω ωστόσο κύριε Πρόεδρε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιμείνει στην διάρκεια των τελευταίων τριών ετών να λαμβάνει την πολιτική απόφαση να αυξάνει τον προπολογισμό του οργανισμού Frontex για να μεταφέρει έτσι, να, δώσει έτσι ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιθυμεί την ενίσχυση του οργανισμού αυτού. Εάν αλλάξουμε την στάση αυτή και αν στη γνωμοδότησή μας πούμε για πρώτη φορά ότι θέλουμε να παραμείνει ο λογαριασμός, συγγνώμη, ο προϋπολογισμός στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, φοβούμε ότι τότε αντιφάσκουμε με το πολιτικό μήνυμα που έχει δώσει το Κοινοβούλιο τα τελευταία τρία χρόνια. Εγώ θα προτιμούσα να μην πούμε τίποτε στην γνωμοδότηση, αντί να πούμε ότι ο προπολογισμό θα πρέπει να παραμείνει στο, στα ίδια επίπεδα με τα περσινά. Έστω και αν αυτό θέλουμε εν τέλει να κάνουμε. Αυτά σε σχέση με την Frontex. Δεύτερο και τελευταίο για την γνωμοδότηση. Θα ήθελα να προσθέσουμε μια παραπομπή για τον μηχανισμό αλληλεγγύης που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όπου ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν θέλουμε απλώς τον μηχανισμό αλληλεγγύης, αλλά ότι χρειαζόμαστε και τους χρηματοδοτικούς πόρους για τον μηχανισμό αυτό. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες του προϋπολογισμού, ως πολιτική ομάδα δεχόμαστε τις περισσότερες από αυτές που έχουν ήδη κατατεθεί, από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, όπου διαφέρουμε διαλόγους αρχής. Θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα όλες οι πολιτικές ομάδες αύριο έγκαιρα πριν από την ψηφοφορία να επιτύχουν συμβασμούς επί όλων των τροπολογιών. Νομίζω ότι αυτό είναι δυνατόν. Εμείς πάντως είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και επιθυμούμε και οι δικές μας τροπολογίες να επιτύχουν την υποστήριξη των άλλων ομάδων. Άλλα σχόλια, ρωτά ο Πρόεδρος. Όπως είπα πριν, έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ορισμένα θέματα. Ίσως αυτό να είναι χρήσιμο. Στέφανη Χάρντ είναι παρούσα. Χαίρετε κυρίε και κύριοι. Δεν είμαι βεβαία ότι τα έχω σημειώσει όλα με την σωστή σειρά. Πάντως αρχίζω με την Frontex. που είναι σημαντικό ε, θέμα και για τους οργανισμούς. Ο προϋπολογισμός της Frontex για το 2010 φτιάχτηκε έχοντας υπόψη την δυνατότητα απορρόφησης της Frontex και νομίζω ότι ο προϋπολογισμός ανταποκρίνεται τα κριτήρια αυτά. Το 2009-2008 υπήρχε κάποια δυνατότητα πρόφησης για πιστώσεις πληρωμών από πλευράς Frontex. Γι' αυτό δεν προτείνουμε εμείς αύξηση των πιστώσεων πληρωμής, διότι υπό τους νέους δημοσιονομικούς κανονισμούς οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τα χρήματα που δεν δαπάνησαν. Και εκτός από αυτό περιοριζόμαστε και από τη δημοσιονομική προοπτική η οποία ε, συμπιέζει τα ανώτατα ποσά. Επί του παρόντος αυτή είναι η άποψή μας. Και όπως είπα, ο προπολογισμό που προτείνει η Κομισιόν είναι αυτός που θεωρούμε ότι είναι ο σωστός. Και η Frontex η ίδια συμφωνεί. Για τις άλλες τροπολογίες η Κομισιόν δέχεται ιδιαίτερα τις τροπολογίες που αναφέρονται στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων με μια μικρή αύξηση της χρηματοδοτησής του διότι υπάρχουν κάποιες πρόσφατες πρωτοβουλίες της Κομισιόν για εσωτερικές ανακατανομές για, την αυξανόμενη, για τις αυξανόμενες αιτήσει δηλαδή που λαμβάνουμε για κονδύλια που θα χρειαστεί να αυξηθούν σημαντικά το 2010. Άλλη τροπολογία που δεχόμαστε είναι η υποστήριξη για μια ιστοσελίδα για τις προξενικές θεωρήσεις και η Κομισιόν ε, θα αναλάβει την πρωτοβουλία αυτή. Οι υπηρεσίες δε της Κομισιόν υποστηρίζουν την ιδέα. Και σε ό,τι αφορά τα ταμεία επιστροφής και άλλα, περιλαμβάνονται ήδη στις τρέχουσες δραστηριότητε μας και δεν χρειάζεται μάλλον να, να προσθεθούν και άλλοι περιορισμοί ή απαιτήσει για την εφαρμογή του το 2010. παρόμοια είναι η άποψή μας και για τις άλλες τροπολογίες που έχουν σχέση με την εγκληματικότητα, με τα ναρκωτικά, με προγράμματα πρόληψης της εγκληματικότητας ή του εγκλήματος που περιλαμβάνονται ήδη στα προγράμματα εργασιών για το 2010. και που ήδη σχεδιάζονται ώστε να ξεκινήσουν στις αρχές του 2010. Αυτά έχουν ενταχθεί στα σχέδιά μας. Είναι επαρκής οι απαντήσεις μου. Ναι, σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας, κυρία εκπρόσωπε της Κομισιόν. Αλλά είδα κάποιο άλλο χέρι να σηκώνεται. Ναι. Αλφάνο, Ταβάρες. Θα επιστρέψω μετά στον κύριο Μπουσούτη. Και μετά θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Κύριος Αλφάνο. Η κυρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξετε τις τροπολογίες Κροτσέτα. Δεν είναι παρόν ο βουλευτής. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο απειλείται από τη μαφία στην Ιταλία κινδυνεύει η ζωή του και δεν είναι εδώ γιατί δεν του δόθηκε η δυνατότητα να έχει την αστυνομική συνοδεία που απαιτείται. Η τροπολογία του ζητά να υποστηριχθούν ορισμένες οργανώσεις και συνεταιρισμοί που διαχειρίζονται τα αγαθά τα οποία έχουν δημευθεί από τη μαφία. Όλες αυτές είναι δραστηριότητες πάρα πολύ σημαντικές ψυχολογικά για τη χώρα μου. Και προτείνει την υποστήριξη επίσης και την ένταξη των μεταναστών στις περιοχές του Νότου. Όλα αυτά πρέπει να υποστηριχθούν από την Επιτροπή μας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ταβάρες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να τονίσω ότι είναι αναγκαίο όποια αύξηση γίνει ή για πολιτικές ή για άλλους οργανισμούς τύπου Frontec να έχουν σχέση άμεση με συγκεκριμένες ανάγκες των οργανισμών αυτών και θα θέλαμε να μας υποβάλουν οι οργανισμοί αυτοί σχέδια λεπτομερή των ενεργειών που θέλουν να αναλάβουν. Κάτι το οποίο το είχαμε της και στο παρελθόν και πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς ε, χρειάζονται για να μην αυξάνονται τα κονδύλια που τους δίδονται για λόγους ε, συμβολικούς ή ε, αλλά για συγκεκριμένες δράσεις και να έχουμε και τα αποτελέσματα της χρησιμοποίησης των κονδυλίων που τους είχαμε χορηγήσει και στο παρελθόν. Μπουσούτιλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, κυρίως για το Frontex. Εδώ και δύο χρόνια διπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό συνολικά της υπηρεσίας αυτής. Όταν πήραμε την πρωτοβουλία Προσπάθησε να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν ήταν αυτό ε, απαραίτητο λόγω της δυνατότητας απορρόφησης. Σέβομαι τις τεχνικές συμβουλές τις οποίες μας δίδει η Επιτροπή, αλλά πήραμε την πολιτική απόφαση να προχωρήσουμε. Όταν πήραμε την πολιτική απόφαση, τότε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο συμφώνησαν μαζί μας. Για το Frontex αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το πολιτικό leadership. Καθυστερήσαμε, ξεκινήσαμε μια προσπάθεια, δεν πρέπει να την εγκαταλείψουμε τώρα. Σχετικά τώρα με τις τροπολογίες οι οποίες ήδη περιλαμβάνονται σε, υπάρχους, σε υπάρχοντες κανονισμούς. Αν οι τροπολογίες αυτές προβλέπονται στον υπάρχοντα κανονισμό, τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη συγκεκριμένη τροπολογία και αυτό το οποίο λέγεται στις τροπολογίες πρέπει να γίνει αυτόματα δεκτό. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό που είπε η Επιτροπή είναι λόγος για την αποδοχή των τροπολογιών και όχι για να αγνοηθούν οι τροπολογίες. Το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια πολιτική υπογράμμιση του σημαντικού στη συγκεκριμένη περίπτωση και να μην αγνοηθεί παρακαλώ η πολιτική μας βούληση. Yes. Uh, we have been uh, carefully listening and... Uh, Προσέξαμε αυτά τα οποία είπατε και σημειώσαμε όλες τις παρατηρήσεις, τις λάβαμε υπόψη και από σας κύριε Αλφάνο και από τον κύριο Ταβάρης και επίσης σημειώνουμε και αυτό το οποίο είπε ο κύριος ε, Μπούσετιλ για τα θέματα του Frontex. συμφωνώ με αυτά τα οποία είπατε και εγώ έχω θέσει ένα αντίστοιχο θέμα όταν, για το Frontex όταν συνέτασα την έκθεση αυτή και συνειδητοποιώ πόσο έχει αυξηθεί ε, η δημοσιονομική κάλυψη των αναγκών του Frontex αλλά είναι απόλυτα φυσιολογικό βέβαια γιατί η διάρκεια ζωής του Frontex μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ μικρή. Πριν λίγα χρόνια όταν εγώ ήμουν υπουργό δικαιοσύνη στην Ισπανική κυβέρνηση, τότε υιοθετήθηκε η απόφαση για το Frontex και μέσα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα έχει πολλαπλασιάσει τους πόρους που έχει στη διάθεσή του. Τίθεται λοιπόν το θέμα το οποίο θέσατε κι εσείς και μου είπαν οι υπηρεσίες με τις οποίες ήρθα σε επαφή ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το Frontex για πρώτη φορά δεν στάθηκε ικανό να φέρει εις πέρας, να εφαρμόσει και να δαπανίσει θα έλεγα τους σπόρους οι οποίοι του είχαν δοθεί. για το συγκεκριμένη θέση του προϋπολογισμού. Πάντως, συμφωνώ με τη λογική την οποία εκφράζεται και προτείνω να προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα έτσι ώστε να βελτιώσουμε την διατύπωση της παραγράφου στην, πρόταση γνωμοδότησής μου. Συμφωνούμε νομίζω επί της ουσίας και θα συνεργαστούμε για την τελική διατύπωση μέσω των υπηρεσιών μας. Όλοι γνωρίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με τη ρήτρα σταθερότητας, εάν αυξήσουμε τους πόρους προς ένα όργανο, προς ένα μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιος άλλος θα πληρώσει το τίμημα, κάποιος άλλος θα επηρεαστεί αρνητικά. Πρέπει όμως να συνεργαστούμε και να δούμε ποια είναι τα προβλήματα, γιατί πράγματι είναι τεράστιο το πολιτικό μήνυμα που στέλνουμε μέσω του Frontex, μέσω της ενίσχυσής του. Και θα πρέπει να συνεχίσετε να αυξάνετε το προπολογισμό του Frontex και όχι να μειούτε. discussion Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να μην καθυστερήσουμε άλλο. Η προθεσμία είναι η 7η Σεπτεμβρίου και μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε καταλήξει σε συμφωνία για να υπάρξει μια πραγματική συνένεση για τις δημοσιονομικές γραμμές ε, για το Frontex. Ε, θα πρέπει να γίνουν δύο ψηφοφορίες. Η μία αφορά την πρόταση για γνωμοδότηση και οι άλλοι τις γραμμές του προϋπολογισμού. Πρέπει να φανούμε, θα έλεγα, γρήγοροι, ταχείς. Θα πρέπει να στείλουμε το μήνυμα το οποίο απαιτείται. Πράγματι ο καθένας από εσά εκφράζει την ευαισθησία της πολιτικής του ομάδας για συγκεκριμένα θέματα. Και σχετικά με το Frontex, πράγματι έχει γίνει ένα βήμα προς τα εμπρός από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε παρά να το υπογραμμίσουμε. Κύριος Ταβάρες, πάλι, μία σύντομη παρέμβαση. Να πω ότι προφανώς και στοχεύουμε στη βελτίωση της τελικής διατύπωσης, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην στέλνουμε πολιτικά μηνύματα με χρήματα χωρίς την απαραίτητη πολιτική γλώσσα, πολιτική ορολογία. Η βελτίωση λοιπόν της τελικής διατύπωσης σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύψουμε τις ανησυχίες που έχουν πολύ σχετικά με το Frontex. Θα πρέπει να δώσουμε τον σωστό πολιτικό προσανατολισμό στο Frontex. Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα στο Frontex αν πράγματι δεν έχει τη δυνατότητα να τα δαπανίσει τα χρήματα αυτά. Αυτό δεν έχει κανένα νόημα και σε επίπεδο φυσικά πολιτικό και σε επίπεδο δημοσιονομικό. Συμφωνούμε όλοι με αυτό. Επαναλαμβάνω ότι το Frontex όμως πριν λίγα χρόνια δεν υπάρχει και τώρα κάνει μια πραγματική δουλειά. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ισπανία, στη Μάλτα. Τα πράγματα αλλάζουν κάπως. Φυσικά το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, ούτε πρόκειται να υπάρχει μια συνεχής αύξηση. Το θέμα είναι όμως να βοηθάμε οικονομικά κάποια όργανα τα οποία έχουν αυτή την ανάγκη γιατί είναι χρήσιμα. Η συζήτηση θα συνεχιστεί εν πάση περιπτώσει εφόσον συμφωνεί και ο κύριος Μπουσούτιλ. Περνάμε στο επόμενο θέμα, παρακαλώ. Με ενημερώνουν ότι η Σουηδική Προεδρία δεν είναι πλέον παρούσα. Α, όχι, είναι παρούσα. Είναι εκεί πίσω. Οπότε έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε το θέμα αυτό της ημερήσια διάταξης. Ο κύριος Κοέλιο, ο οποίος θα έπρεπε να παρουσιάσει τα σημεία 8 και 9, ή μάλλον 9 και 10, ο κύριος Κοέλιο δεν είναι παρόν. Προς το παρόν, μπορεί να έρθει αργότερα. Α, όχι, θα συζητηθεί στην επόμενη τακτική συνάντησή μας το τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Νομίζω όμως ότι έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, έτσι ώστε να καλύψουμε τον χρόνο μας μέχρι τις 6.30. Παρακαλώ την εκπρόσωπο της Προεδρίας να έρθει εδώ και να ακούσουμε τις απόψεις της Προεδρίας για τη σωματεμπορία. We invite again the Swedish presidency on human trafficking and then... Λοιπόν, έχετε το λόγο, αλλά σας θυμίζω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο βέβαια, γιατί νομίζω ότι στις 6.30 σε 15 λεπτά από τώρα θα κλείσει η συνεδρίαση och eh, tacka Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα εκλεκτά μέλη. Θα είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Λίγα λόγια θα πω μόνο. για τις δράσεις τις οποίες προτείνουμε για την καταπολέμηση της σώματεμπορίας από την ε, Σουηδική Προεδρία. Και θα δώσω το λόγο και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας μιλήσει για την υποσυζήτηση απόφαση πλαίσιο. Όπως είπε και ο Υπουργός, ή Υπουργός μάλλον σήμερα το πρωί, η καταπολέμηση του φαινομένου αυτού είναι κάτι το καθοριστικό για τη Σουηδική Προεδρία. Εμείς προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας στην καταπολέμηση των πηγών θα έλεγα που παρέχουν το υλικό σε εισαγωγικά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας με τις τρίτες χώρες. Και κάθε χώρα με την οποία συζητάμε, με τα Δυτικά Βαλκάνια, με τις Ηνωμένε Πολιτείες, με τη Ρωσία κτλ. Τίθεται το θέμα στον τομέα ο οποίος μας Μας ενδιαφέρει έχουμε σαν στόχο να διαμορφώσουμε μια σαφή στάση θα έλεγα η οποία να είναι μια σταθερά, να αποτελεί μια σταθερά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια των διεθνών προσπαθειών εκρίζωσης του φαινομένου αυτού. πιο συγκεκριμένα προτείνουμε ένα πρόγραμμα δράσης, ένα έγγραφο στρατηγικής. Δεν θα μπω τώρα στις ε, προτάσεις στο σύνολό τους γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα υπάρξει μια συνάντηση και με τις τρίτες χώρες στις 19 και 20 Οκτωβρίου. Θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα σε εκπροσώπους Υπουργείων και από τη ΣΥΠΑ και τη Ρωσία και θα δώσω αμέσως τώρα πια το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Σκορμπίνσκι. Ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορούμε να συζητήσουμε για πρώτη φορά στα πλαίσια του νέου κοινοβουλίου το θέμα αυτό της σωματεμπορίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφό της του προηγούμενου Οκτωβρίου λέγει ότι ο αριθμός των ανθρώπων που εισάγονται σε εισαγωγικά στην Ευρώπη για τέτοιους παράνομους λόγους είναι εκατοντάδες χιλιάδες ενώ οι δικαστικές διαδικασίες, οι, οποίες, οι ποινικές διαδικασίες οι οποίες ξεκίνησαν πέρυσι δεν ξεπερνούσαν τις εκατό. Αυτό είναι κάτι το φοβερό. Γι' αυτό και προτείναμε να υπάρξει ένα νέο πλαίσιο καταπολέμησης του φαινομένου. Αυτό τη συμφωνία πλαίσιο, η απόφαση πλαίσιο, προτείνει μια στρατηγική αντιμετώπιση του φαινομένου που συνδυάζει τη δίωξη των παρανόμων, την προστασία των θυμάτων και την περαιτέρω πρόληψη του φαινομένου στην πηγή. Οι ξεκίνησαν, οι συζητήσεις ξεκίνησαν τον Απρίλιο στο Συμβούλιο και σας ενημέρωσε γύρω από αυτό ο εκπρόσωπος της Σουηδικής Προεδρίας. Να σας πω λίγα από τα βασικά στοιχεία των προτάσεων της Επιτροπής. Υψηλότερες ποινές, επιβαρυντικές συνθήκες, στρέφουμε την προσοχή μας στα θύματα, αποτρέπουμε την τιμωρία και της κυρώσεις εις βάρος των θυμάτων, φυσικά ιδιαίτερα των παιδιών όταν απλά καταδικάζονται για μικρές κλοπές. Τίθεται το θέμα των δικαστικών δικαιοδοσιών, έτσι ώστε να μην γλιτώνουν οι παράνομοι και να θεωρείται το θέμα αυτό σαν ένα σοβαρό έγκλημα σε όλες τις χώρες, κάτι το οποίο να σημαίνει και τη δυνατότητα χρήσης όλων των μέσων και των μεθόδων. Επαναλαμβάνω στα πλαίσια της αντιμετώπισης του θύματος στο κέντρο της προσπάθειας την οποία κάνουμε, εισάγουμε κάποια μέτρα τα οποία έχουν σαν στόχο την θυματοποίηση, την αποφυγή της θυματοποίησης των θυμάτων, έτσι ώστε τα θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης να μην είναι υποχρεωμένα κατά τη διάρκεια της δίκης να αντιμετωπίζουν τους διώκτες τους. Επίσης προτείνουμε και μέτρα υποστήριξης των θυμάτων, να δώσουμε την δυνατότητα στα θύματα αυτά, εφόσον το επιθυμούν, να συνεργαστούν με τις ανακριτικές αρχές. Κάτι το οποίο σε ορισμένες χώρες έχει παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο. Σε επίπεδο πρόληψης, προσπαθούμε να δούμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για τη μείωση της ζήτησης στη σωματεμπορία. Εμπνεώμεθα και από το Ολλανδικό παράδειγμα, και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να, να ορίσουν εθνικούς εισηγητές με ομόλογους μηχανισμούς σε κάθε χώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε σωστά την εφαρμογή των πολιτικών αυτών. Όπως ξέρετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη εγκληματική δραστηριότητα για να την εντοπίσει κανείς και απαιτείται να υπάρξει μια εξαιρετική μορφή συνεργασίας πολλών υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνίας των πολιτών, γραφείων εργασίας, διοκτικών αρχών κτλ. Αν δεν υπάρξει συνεργασία αυτή τότε δεν υπάρχουν δυνατότητες σωστής δίωξης. Ευχαριστούμε τη Σουηδική Προεδρία γιατί προχωρά προς τη σωστή κατεύθυνση και δίνω το λόγο τώρα στην συνάδελφο Πινελόπη. Πάρα πολύ σύντομα θα πω το εξή. Η πρόταση έγινε αποδεκτή θετικά. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τα φαινόμενα σε υψηλό επίπεδο. Η προσοχή μας mm. εστιάζεται στο εξής. Θα πρέπει να βρούμε νέα στοιχεία που θα συνδυάσουμε με τις ε, παραδοσιακές νομοθετικές πράξεις για να βοηθηθούμε και να προχωρήσουμε. Ήδη το πρόθεσε αρκετά το θέμα η Τσεχική Προεδρία και εμεί συνεχίζουμε με την ίδια ταχύτητα. Το πνεύμα μας είναι δημιουργικό και δυναμικό, ενεργητικό. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια ε, θέματα πιο δύσκολα από άλλα. Ο Γιάκομπ ε, σας ανέφερε κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν και αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης, δεδομένου ότι έχουμε διαφορετικά ε, νομοθετικά συστήματα τα οποία πρέπει να προσπαθήσουμε να συντονίσουμε. Κάποιο άλλο θέμα επίσης το οποίο χρειάζεται χρόνο μελέτης είναι να δούμε πώς θα εφαρμοστεί το σύνολο των ποινικών κυρώσεων θα επιβληθούν, δηλαδή το ποινικό δίκαιο γενικότερα. Δεδομένου ότι υπάρχουν απάτες, υπάρχουν πιέσεις, Πολλές φορές ε, ε, υφίστανται πιέσεις ε, τα θύματα για να συνεχίσουν να έχουν παραβατική συμπεριφορά ή να εγκληματούν και όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα εξετάσουμε έγκαιρα. Ευχαριστώ σας, ευχαριστώ και εκτιμούμε την σύντομη παρουσίαση που έκαναν οι διάφοροι πρόσωποι της Σουηδικής Προεδρίας για το τόσο σημαντικό θέμα αυτό που είναι η σωματεμπορία. Όπως ξέρετε, οι διερμηνείς ε, εργάζονται κάποιες συγκεκριμένες ώρες. Ζητώ την κατανόησή σας. Δεν μπορούν να ξεπερνούν πάντα την ώρα τους. Σήμερα Είχαμε μία πάρα πολύ φορτωμένη μέρα. Κάναμε πολύ σημαντικές συζητήσεις για θέματα ουσίας. Και επειδή είναι αργά, θα ήθελα για τη συζήτηση να πω το εξής. Να υποβληθούν γραπτός τα ερωτήματα στην Κομισιόν και στην Σουηδική Προεδρία που είμαι σίγουρος ότι ευχαρίστως θα σας αποστείλουν και γραπτό τις απαντήσεις τους. Σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα στην επόμενη συνεδρίαση της ε, Επιτροπής μας προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, συγκεκριμένα στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου. Νομίζω ότι όλοι σήμερα αρκετά εργαστήκαμε. Θα διακόψουμε τις εργασίες μας και θα σας ξαναδώ όλους αύριο στις 9 το πρωί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.